Uh, αγαπητοί συναδελφοί, θα ήθελα να σας ζητήσω να καθίσετε παρακαλώ, διότι θα ξεκινήσουμε αμέσως. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά σας για να παρακολουθήσετε τη συζήτηση στη μητρική σας γλώσσα. Θα ήθελα καταρχήν να σας ευχαριστήσω για τις χθεσινές συζητήσεις και τις συναντήσεις διότι όπως γνωρίζετε οι εισηγητές των ομάδων εργασίας ε, θα κάνουν αμέσως τώρα τις παρουσιάσεις ε, των πορισμάτων. Καταρχήν όμως θα ήθελα να σας ε, πληροφορήσω ότι η Προεδρία των, του Κοινοβουλίου και της Γερουσίας της ε, Ισπανίας αποσιάζουν σήμερα διότι η Ισπανική κυβέρνηση λαμβάνει σήμερα πολύ σοβαρές αποφάσεις και στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε κατανόηση ε, γι' αυτό διότι αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει μία δύσκολη κατάσταση γι' αυτό ο και οι πρόεδροι του Κοινοβουλίου και της Γερουσίας της Ισπανίας πρέπει να βρίσκονται επί τόπου και το κατανοούμε. Θέλω όμως να καλωσορίσω τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Γιώργη Μαλμούνια, ο οποίος θα μας μιλήσει και θα ακούσουμε τα σχόλιά του με πολύ ενδιαφέρον ο κύριος Πέντρο Μαρίν Λουίς Ορίμπα που εκπροσωπεί την ε, Ισπανική Προεδρία την εναλλασσόμενη η οποία είναι ε, πολύ ε, σημαν... εναλλασσόμενη Προεδρία της Ευρώπης και αυτό είναι πολύ σημαντικό όπως ξέρετε για το νομοθετικό μας έργο διότι η εναλλασσόμενη Προεδρία αυτή τη στιγμή είναι ε, στην Ισπανία και ε, ο εκπρόσωπος της Ισπανικής Προεδρίας θα μπορέσει επίσης να λάβει το λόγο και μπορούμε να του απευθύνουμε ερωτήσεις εάν χρειαστεί. Θα ήθελα με αυτή την ευκαιρία να σας πω ότι από την αρχή ότι οι κοινοβουλευτικές μας υπηρεσίες έχουν ε, συμβάλει πολύ σε αυτή τη συνεδρίαση και η κυρία Μπέργκερ η οποία είναι διευθύντρια του κέντρου μας για την οργάνωση αυτών των συνεδριάσεων και ο κύριος Μπερνάτσκι ο οποίος είναι επικεφαλής των ομάδων εργασίας και προετοίμασαν αυτή τη συνεδρίαση αξίζουν τις ευχαριστίες όλων μας ε, για την οργάνωση αυτών των συνεδριάσεων όπως άλλωστε και η Ισπανική Προεδρία, η Ισπανική Κυβέρνηση οι οποίες ε, συνέβαλαν ε, σημαντικά και γι' αυτό μπορέσαμε να επωφεληθούμε της βοηθείας τους. Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω όλους αυτούς οι οποίοι συνέβαλαν στο να εξελιχθούν ομαλά οι εργασίες μας. Τώρα όμως προχωρούμε στη συζήτηση και θα ξεκινήσουν οι παρουσιάσεις των εισηγητών μας. Θα ήθελα λοιπόν να ζητήσω από τους ε, εισηγητές ε, να τηρήσουν δεκάλεπτα το παρουσίασης ε, και ξεκινώ με τον κύριο Σάιρους Βόλσκι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ο οποίος θα λάβει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θέλω να σας παρουσιάσω τα αποτελέσματα της πρώτης ε, ομάδος ε, εργασίας σχετικά με την ασφάλεια ε, και την ποικιλία παροχής ενεργείας. Ε, βασιστήκαμε στο άρθρο 194 της συνθήκης το οποίο θα πρέπει να βελτιωθεί για να μπορέσουμε να μιλάμε με μία φωνή ε, και πρέπει να εξετάσουμε τα θέματα αυτά στα πλαίσια της συνεργασίας και με τα γεωπολιτικά θέματα και την ασφάλεια διότι είδαμε χθε ότι έχει βελτιωθεί η συνείδηση των ε, θεμάτων ενεργειακής ασφάλειας στα κοινοβούλια κοινοβούλια της Ευρώπης και ε, στις συζητήσεις μεταξύ εθνικών βουλευτών και ευρωβουλευτών. Ε, ε, την περίοδο των κρίσεων διαπιστώσαμε ότι τα κράτη-μέλη δεν μπορούσαν να αντιδράσουν ικανοποιητικά ή επαρκώς στις κρίσεις αυτές. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια πιο συντονισμένη κίνηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο και μια πολιτική ευρωπαϊκή η οποία θα είναι εξοπλισμένοι με τα αναγκαία μέτρα. Το, η δοκιμασία για την ε, ασφάλεια αυτή ε, είναι προημών, δηλαδή ε, συζητιέται με το Συμβούλιο και θα πρέπει να μπορούν τα κράτη-μέλη να καταρτίζουν το σύστημά τους παροχής σε βάση του άρθρου 194 της Θα πρέπει να υπάρχει όμως μια ευρωπαϊκή πολιτική ανάλογη της προκλήσεως με τα αναγκαία πολιτικά και νομοθετικά μέτρα. Ε, τα συμπεράσματα της πρώτης ομάδος εργασίας εχθές είναι τα εξής. Ε, ε, συμφωνήσαμε ότι ενώ υπάρχουν νομοθετικά εργαλεία δεν έχουν εφαρμοστεί επαρκώς λόγω ελήψεως πολιτικής θέλησης και μακροπρόθεσης και ε, και μακροπρόθεσμου οράματο ε, Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε αυτά ήταν πιο φιλόδοξο από ότι η Επιτροπή, το Συμβούλιο και τα κράτη-μέλη. Ζητήσαμε ε, να υπάρξει επέμβαση σε ορισμένες καταστάσεις διότι οι μηχανισμοί της αγοράς είναι το πρώτο μέσο για να καταπολεμήσει κανείς τις διαταράξεις της παροχής αλλά δεν υπάρχει μία ικανότητα ικανοποιητική ενιαία αγορά ενεργείας εάν δεν είναι εξασφαλισμένος ο χώρος ασφαλείας ενεργειακής παροχής. Στηρίξαμε την αρχή της αλληλεγγύης αλλά τέθηκε το θέμα της χρηματοδοτήσεως της εφαρμογής της και γι' αυτό συμφωνήσαμε ότι θα πρέπει να διατυπωθεί ένα σωστός μηχανισμός σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την ε, ε, κάλυψη της ασφάλισης και της διασύνδεσης. Όσον αφορά την πρόσταση Μπούζεκ Ντελόρ πρέπει να δούμε αν χρειαζόμαστε ε, ένα ή περισσότερα κοινά μέτρα και συμφωνήσαμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να έχει μεγαλύτερη αλληλεγγύη με τη μορφή που έχει και το Σέγγεν στο μέλλον κατά τρόπον ώστε να μην βασιζόμαστε μόνο στην ε, ομάδα ε, και το πουλ που έχει δημιουργηθεί για την κάλυψη των αναγκών. Όσον αφορά την ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή Τη της έναντι τρίτων χωρών αναφορά με τα παραδείγματα της Λευκορωσίας και Ουκρανίας οι οποίες πιέζονται και τονίσαμε ότι το αέριο δεν είναι μόνο μία πρώτη ύλη αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν πολιτικό μέσο για να εμποδίσει την ε, Ευρώπη να έχει μία κυρίαρχη ενεργειακή πολιτική. Όσον αφορά την Τουρκία, ε, αγωγός Ναμπούκο είναι πολύ σημαντικός και τονίστηκε ότι η Άγκυρα πρέπει να συνεργαστεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς να συνδέει όμως τα δύο θέματα αυτά διότι δεν ε, έχει σχέση η ενεργειακή παροχή με τις διαδικασίες προσχωρήσεως της Τουρκίας. Θα έπρεπε ε, επίσης ε, να εξασφαλίσουμε εναλλακτικέ πηγές ενεργείας για να μπορέσουμε να αντιβεξέλθουμε τις κρίσεις διότι ε, βλέπουμε ότι τώρα υπάρχουν πολύ μεγαλύτερες ανάγκες π.χ. φυσικού αερίου από ό,τι στο παρελθόν και μας απέδειξαν οι Βρετανοί φίλοι μας. Συμφωνήσαμε λοιπόν ότι το μείγμα παροχής ενεργείας πρέπει να παραμείνει στη διάκριση των κρατών μελών και να είναι μία λύση για να διαφοροποιήσουν τις λύσεις ε, του παροχής στο μέλλον και να αυξήσουν την ε, ασφάλεια στον τομέα αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χρειάζεται μία μακροπρόθεσμη στρατηγική, περαιτέρω έρευνα και βραχυπρόθεσμα ασφάλεια της παροχής ε, αερίου και πετρελαίου πετρελαίου γι' αυτό και πρέπει να επιτύχουμε έναν όσο δυνατό πιο φιλόδοξο συμβιβασμό για την ρύθμιση ε, της παροχής αερίου που διαπραγματεύεται τώρα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με το Συμβούλιο ε, διότι υπάρχει μια φιλόδοξη ε, προσέγγιση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την οποία στήριξαν οι περισσότεροι συνάδελφοι από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την έκθεσή σας. Και εν ονόματι όλη της πρώτες ομάδες εργασίας ευχαριστώ τους συναδέλφους για την εργασία τους. Τώρα η ομάδα εργασίας 2. Ο κύριος Φέλιξ Λαβίλα Μαρτίνες από την Ισπανία έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Αντιπρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, κύριε Υφυπουργέ, κύριοι βουλευτές, ε, ευρωβουλευτές, ε, για την έκθεση της ομάδας μας όσον αφορά τα θέματα ενέργειας μετά από έντονες εργασίες στο, στους κύκλους της Επιτροπής. Χωρίς ενιαία αγορά ενέργειας δεν θα υπάρξει η Ευρωπαϊκή Κοινότητα στα ενεργειακά θέματα στον 21ο αιώνα. Για να υπάρξει όμω μια τέτοια αγορά και να υπάρξει ανταγωνισμό με βάση πιο ανταγωνιστικά τιμολόγια, με τη διασφάλιση του ανεφοδιασμού και αηφορία, θα πρέπει να είναι διασυνδεδεμένα τα ηλεκτρικά δίκτυα. Χωρί διασύνδεση των ηλεκτρικών δικτύων και του φυσικού αερίου δεν θα υπάρξει ενιαία αγορά και δεν θα μπορέσει να είναι ανταγωνιστική η Ευρωπαϊκή Ένωση στον 21ο αιώνα. Υπήρξε απόλυτη συμφωνία στην ομάδα εργασία στον κατεπήγοντα χαρακτήρα να πετύχουμε αυτό το στόχο και να βελτιστοποιήσουμε αυτή την πτυχή. Και θα πρέπει να δραχθούμε του νομικού πλαισίου που έχουμε στη διάθεσή μα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιαίτερα μετά την έναρξη σε ισχύ τη συνθήκη Λισαβόνα. Αυτή τη στιγμή αυτή η διασύνδεση ενεργειακή στο κοινοτικό επίπεδο δεν υφίσταται και χρειάζεται η μέγιστη πολιτική προώθηση Επίσης, οι στόχοι της διασύνδεσης που καθορίστηκαν στην Ευρωπαϊκή Σύνοδο το 2002 στη Βαρκελόνη δεν υλοποιήθηκαν. Οι Ευρωπαίοι πολίτες ε, και η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων απαιτούν κατεπίγουσες λύσεις, βελτιώνοντας επίσης την αποτελεσματικότητα εξοικονομώντας ε, ενέργεια με την βέλτιστη δράση στην ε, μεταφορά ακόμα και με ηλεκτρικά οχήματα. Υπογραμμίσαμε ότι αν δεν λάβει αποφάσεις και μάλιστα κατεπηγόντως η Ευρώπη και με συντονισμένο τρόπο κάθε φορά θα μετράμε λιγότερο στον παγκόσμιο, ε, θα έλεγα, στην παγκόσμια σκηνή. Μια ενιαία αγορά ενέργειας ε, με διασυνδεδεμένα δίκτυα από πλευράς ευρωπαϊκών χωρών θα μπορέσει να προωθήσει την καινοτομία στις ε, ανανεώσιμες και αηφόρες πηγές ενέργειας. Θα δημιουργήσει δυνατότητες απασχόλησης και θα μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να δημιουργήσει το επίπεδο ευημερία. Μια αγορά ενέργειας είναι πιο αηφόρα με διασυνδεδεμένα δίκτυα στην Ευρώπη. Επιπλέον, δρατώμενη της ευκαιρίας για την καινοτομία θα μπορέσει να λειτουργήσει ο ανταγωνισμός και η ασφάλεια ανεφοδιασμού. Η Ευρώπη θα είναι περισσότερο Ευρώπη για τους πολίτες όταν θα λύνει προβλήματα συγκεκριμένα, με συγκεκριμένο τρόπο. Δεν έχει σύνορα η ενέργεια και πρέπει να εξυπηρετήσει τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να αποφύγουμε προβλήματα στον ανεφοδιασμό όπως αυτά που ζήσαμε η αγορά δεν ήταν η ίδια σε θέση να δημιουργήσει αυτή τη δυνατότητα μεταφοράς. Θα πρέπει να προωθήσουμε τη διαλειτουργικότητα και τις μεταφορές. Γι' αυτό χρειάζεται κρατική χρηματοδότηση, δημόσια χρηματοδότηση. Η ενέργεια έχει άμεση επίπτωση στις τιμές και στον πληθωρισμό. Πρέπει να βελτιώσουμε την εξοικονόμηση και να είμαστε πιο ανταγωνιστικοί. Μια οικονομία που θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για να παράγει τα ίδια προϊόντα θα είναι πιο ανταγωνιστική και πιο αηφόρα υποδείξαμε το τι πρέπει να γίνει. Επιμείναμε στο ότι η τεχνολογική ανάπτυξη και η αγορά θα πρέπει να καθορίζουν τις εξελίξεις. Σχολιάστηκε και είπαμε ότι ο άνθρακας είναι μια σταθερή πηγή ενέργειας. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τις ε, καινοτομίες ε, τις τεχνολογικές και με τη σύλληψη του διοξιδίου του άνθρακα μπορούμε να μειώσουμε την εξάρτησή μας ε, από ενεργειακά προϊόντα. Αναφέρθηκε η ανάγκη επίσης να προωθήσουμε μέτρα για να ε, αντισταθμίσουμε ε, την κατάσταση σε σχέση με το πετρέλαιο. Κάτι όμως το οποίο δεν έχει γίνει πλήρως. Υπήρξε απόλυτη συμφωνία και συνένεση να προστατέψουμε περισσότερο τους καταναλωτές, με πιο προσιτές τιμές, με πιο καθαρή ενέργεια, σε μια ενιαία αγορά με μεγαλύτερη απελευθέρωση. Σύμφωνα με την, τις οργανώσεις του ΟΗΕ έχουμε πάμπολους που δεν έχουν στη διάθεσή τους ηλεκτρική ενέργεια. Πρέπει να συνεισφέρει η Ευρώπη να επιληθεί το πρόβλημα, προωθώντας καθαρές πηγές ενέργειας, επιπλέον έχοντας διπλό όφελος. Θα αποφύγουμε να υπάρξει μεγαλύτερη ρήπανση και θα έχουμε στο μέλλον δεσπόζοντα ρόλο σε αυτές τις αγορές. Ε, ένα τέτοιο παράδειγμα είναι και το παράδειγμα συνεργασίας στη Μεσόγειο. Και επίσης ε, για την ενιαία εσωτερική αγορά θα πρέπει να δούμε ότι με την περίπλοκη αυτή διασύνδεση διαφορετικών ε, σιδηροδρόμων ε, έχουμε προβλήματα να επιλύσουμε. Θα ήθελα να ολοκληρώσω, να με αυτά που είπε ο William Shakespeare, που είναι πολύ κατάλληλο παράθεμα. <clears throat> Ισχυροί λόγοι, είναι, ε, ισχυροί, ε, ισχυροί λόγοι απαιτούν ισχυρέ δράσει. Κυρίε και κύριοι, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να λάβει αυτέ τι στεναρέ δράσει ήδη σήμερα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ συνάδελφε για την παρουσίασή σου. Ευχαριστώ και όλους τους συναδέλφους της ομάδας εργασίας σας οι οποίοι συνεργάστηκαν για ένα δύο χθε το απόγευμα. Ο συνάδελφος Λόπες από την Ισπανία θα μας παρουσιάσει τώρα τα αποτελέσματα των εργασιών της ομάδας εργασίας υπαρίθμου 3. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Αντιπρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κύριε ε, Υπουργέ για θέματα ενέργειας, κυρίες και κύριοι εθνικοί βουλευτές και ευρωβουλευτές. Αυτό που θα κάνω είναι, θα κάνω μια σύνοψη συμπερασμάτων της ομάδας εργασίας υπαριθμών 3 που εργάστηκε χθες το απόγευμα Πρόκειται για την ομάδα ενέργεια και περιβάλλον, ε, νέες μορφές ενέργειας, αηφορία. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συμμετείχαν στην ομάδα εργασίας για την ποιότητα των παρεμβάσεών τους, καθώς και τις ε, συνεισφορές και παρεμβάσεις που καταδεικνύουν σαφή δέσμευση υπέρ της προάσπισης ε, του περιβάλλοντος, ε, του σεβασμού του περιβάλλοντος στο μέλλον ε, το βιομηχανικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την ανάπτυξη καθαρών πηγών ενέργειας και την προαγωγή, την προώθηση αηφόρων πηγών ενέργειας. Ως προς αυτά συζητήσαμε και προβληματιστήκαμε για διαφορετικά θέματα. Πρώτα απ' όλα, υπήρχε σαφή σύμπτωση και συμφωνία ότι οι ενεργειακές πολιτικές είναι προτεραιότητα για την Ευρώπη. Επίσης είναι ένα διαρθρωτικό δομικό στοιχείο, όπου πρέπει σε αυτό να δομήσουμε, να οικοδομήσουμε τη νέα Ευρώπη των πολιτών και των επιχειρήσεων. Γι' αυτό είναι αναγκαίο να επιτύχουμε τους τρεις στόχους, θεμελιώδεις στόχους του Ευρωπαϊκού Ενεργειακού Συστήματος. Πρώτον, ανταγωνισμό. Δεύτερον, ασφάλεια του εφοδιασμού και αηφορία. Για να πετύχουμε αυτούς τους τρεις στόχους στρατηγικού χαρακτήρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη που την συναπαρτίζουν πρέπει να συνεχίσουν το έργο, την εργασία με έντονο ρυθμό, ώστε να υπάρξει μια οικονομική κοινότητα ενεργειακή αποδοτικότητα σε υψηλό βαθμό, αυξάνοντας ε, όσον αφορά την ε, ε, χρήση των ενεργειακών πόρων, βελτιώνοντα την με χαμηλές εκπομπές τρύπων, μειώνοντας την εξάρτησή μα από τρίτους, αυξάνοντα την αποτελεσματικότητά μας σε χρήση με τι ενεργειακέ πηγέ. Εκεί ακριβώ πρέπει να δούμε το θεμελιώδη ρόλο των ανανεώσιμων πηγών ενέργεια και των νέων τεχνολογιών για να πετύχουμε αυτού του τρει στόχου στου οποίου προαναφέρθηκα. Είναι σκληρή δουλειά στην ε, γραμμή την οποία αναπτύσσει και η Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2006 όταν είχαμε το δεσμευτικό στόχο να αυξηθεί το επίπεδο των ε, ανανεώσιμων πηγών ενέργεια από το 7% στα 20% μέχρι το 2020. Σαφή σύμπτωση για να τονίσουμε όσον αφορά αυτά τα εθνικά προγράμματα και σχέδια τα οποία πρέπει να υποβληθούν αυτό τον μήνα του Ιουνίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά δεύτερο λόγο, αναφέρθηκε ότι είναι αναγκαίο να ενισχυθεί η συνεργασία με μια κοινή ενεργειακή αγορά. Και ω προ αυτό είναι θεμελιώδε στα θέματα τη ενέργεια και των καθαρών ε, πηγών ενέργεια να πορευόμαστε προς μια ενιαία κατεύθυνση με μηχανισμούς οικονομικούς και φορολογικούς που είναι αναγκαίοι φυσικά για να διαρθρωθούν και να δομηθούν οι κοινέ αυτές πολιτικές στο εθνικό επίπεδο. Αυτό χρειαζόμαστε ώστε μέσω πρόθεσμα και μακροπρόθεσμα η αηφορία στην τεχνολογία να είναι ο κύριος τομέας που θα δημιουργεί ευημερία σε αυτή τη νέα Ευρώπη. Ω προ αυτό υπήρξε ευρεία συνένεση σε δύο πτυχές. Πρώτον, στο να συνδυάσουμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όχι μόνο με την αηφορία και φυσικά με την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών αλλά και με τον ε, ανεφοδιασμό, την ασφάλεια στον ανεφοδιασμό. Είναι θεμελιώδες να υπάρχει πρόσβαση στα δίκτυα. Δεύτερον, σε ευρωπαϊκή κλίμακα τα εθνικά δίκτυα να είναι επαρκώς διασυνδεδεμένα ώστε να επιτρέπεται η εκμετάλλευση του δυναμικού των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ευρώπη και η βελτιστοποίηση του κόστους των τιμολογίων σε μια αγορά που θα είναι διασυνδεδεμένη. Τρίτον, η προώθηση ευφυών δικτύων. Δεύτερον, ε, ε, ε, ως, ως αυτά πρέπει να υπάρξει η μεγάλη προσπάθεια στις καινοτομίες. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι η ανάπτυξη και οι δράσεις άλλων ε, εμπλεκόμενων στο διεθνές επίπεδο θα πρέπει να μας κάνουν να κινητοποιηθούμε για να μην μείνουμε πίσω. Ως προς αυτό η τεχνολογία πρέπει να επιτρέπει την ανάπτυξη της διασύνδεσης ε, όπως ανέφερα πιο πριν για να διασφαλίζουμε την ε, κάλυψη των ενεργειακών αναγκών και να βρεθούμε στο ύψος των δεσμεύσεών μας. Δεύτερον, οι τεχνολογίες θα πρέπει να συνεισφέρουν στο να μειωθεί το κόστος των ανενώσιμων πηγών ενέργειας και βοηθώντας η Ευρωπαϊκή Βιομηχανία βιομηχανία να βρεθεί στην πρωτοπορία των τεχνολογιών που θα δίνουν τη δυνατότητα να μειώσουμε τις εκπομπές ρήπων θερμοκηπίου και διοξιδίου του άνθρακα και να βελτιώσουμε την επίδοσή μας, την μας, αποδοτικότητά μας στα θέματα ενέργειας. Σημαντική είναι η καινοτομία και η τεχνολογική ανάπτυξη για το ηλεκτρικό όχημα για παράδειγμα, για τα καύσιμα δεύτερης γενναίας ε, που θα βοηθήσουν να μειώσουμε την εξάρτησή μας στα θέματα τα ενεργειακά και θα βελτιώσουν τις εκπομπές ρήπων μειώνοντάς τες, ε, μια και αυτές ρηπαίνουν το περιβάλλον καταλήξαμε στο ότι η πιο αποτελεσματική ενέργεια είναι η ενέργεια εκείνη η οποία δεν καταναλώνεται αλλά αποθηκεύεται και εξοικονομούμε. Έτσι λοιπόν πρέπει να δούμε το θέμα της εξοικονόμησης ενέργειας στο μέλλον. Βασιστήκαμε και τονίσαμε στην ανάπτυξη όχι μόνο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αιωλικής, ηλιακής αλλά και άλλων τεχνολογιών όπως εκείνη που θα προέρχεται από τα απόβλητα, την εκμετάλλευση των αποβλήτων ή και την βιομάζα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Και αυτό το τελευταίο είναι σημαντικό σημαντικό για να διαδραματίσουμε ρόλο στην ε, ανάπτυξη και στην ύπεθρο ε, και λαμβάνοντας υπόψη και τα δάση μας και το περιβάλλον. Επίσης η φορολογία όχι μόνο όσον αφορά την επιβολή φόρων και τελών αλλά και να διευκολύνουμε με φορολογικά κίνητρα τις δράσεις για τις επιχειρήσεις. Να έχουμε και επαρκείς κυρώσεις από την άλλη πλευρά ώστε να έχουμε και αποδοτικότητα στην ε, χρήση της θέρμανσης και της, του κλιματισμού στα κτίρια. Έχουμε την ανάγκη ενός ευφυούς προγράμματος για την ενέργεια και οικονομικούς και δημοσιονομικούς μηχανισμούς για τα κονδύλια που χρειάζονται για να λειτουργήσουν όλα αυτά. Εν τέλει, εν κατακλείδη, τονίσαμε επίσης ότι είναι αναγκαίο να εργαστούμε και να δούμε πέρα από το στενό ορίζοντα τι πρέπει να γίνει μακροπρόθεσμα. Σε σχέση με την ε, μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη ανάπτυξη μέχρι το 2020-2030. Γιατί η καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών απαιτούν μια βιομηχανία πάγια, ισχυρή και ανταγωνιστική. Και θα ολοκλήρωνα λέγοντας ότι είναι μια δέσμευση που έχουμε όσον αφορά τη σημερινή γενναία, τι σημερινέ γενναίες αλλά και τις μελλοντικές γενναίες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ τον Ισπανό συνάδελφο για την παρουσίαση που έκανε σχετικά με τις εργασίες της ομάδας εργασίας Υπερθυντρία. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω συνολικά τους εισηγητές για, ε, για τη συνεργασία τους και για το πνεύμα συνεργασίας το οποίο επέδειξαν όλα τα μέλη των ομάδων εργασίας. Θα δώσω τώρα το λόγο στον εκπρόσωπο του Συμβουλίου, ε, τον κύριο Μαρίν Ουρίμπε. Καλημέρα σας Πρόεδρε, Επίτροπε, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Σας ευχαριστώ πολύ πρώτα απ' όλα που προσκαλέσατε την Ισπανική Προεδρία του Συμβουλίου σε αυτή τη σημαντική συνεδρίαση στην οποία γίνονται συζητήσεις για τα θέματα τα ενεργειακά που είναι ένα θέμα απαραίτητο που πρέπει να εξεταστεί και σε εθνικό επίπεδο και στο επίπεδο τη Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξέρω ότι το θέμα του αν χρειαζόμαστε μια συγκεκριμένη συνθήκη για τα θέματα τη ενέργεια στην Ευρώπη συζητήθηκε χθε και ότι επιπλέον γνωρίζω επίσης, έχω συνειδητοποιήσει ότι έχει συζητηθεί σε, διάφορες, σε διάφορους φορείς αυτό το θέμα. Ο, παρότι ως Προεδρία δεν έχουμε μια θεσμική θέση επ' αυτού, θεωρώ ότι είναι σκόπιμο και μια και τελειώνει ουσιαστικά η περίοδος της Ισπανικής Προεδρίας, να κάνουμε μια επισκόπηση για κάποια θέματα που πιστεύω ότι μπορούν να δώσουν, να ρίξουν φως σε αυτά τα θέματα της συζήτησης. Και θα το κάνω αυτό λαμβάνοντας υπόψη τα βιώματα και τις ευθύνε μου τους τελευταίους μήνες. Ίσως θα μπορούσε να ε, θεωρηθεί μήπως ε, υπό τους σημερινούς όρους και προϋποθέσεις θα έπρεπε να υπάρξει ένα νέο όργανο παρόμοιο με μια νέα συνθήκη ή ένα ε, μέσο το οποίο έχουμε ήδη στη διάθεσή μας αν αυτό θα υπαρκούσε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι η συνθήκη Λισαβόνα ε, άσκησε πρωταγωνιστικό ρόλο και ξεκίνησε με την Ισπανική Προεδρία. Μεταξύ των καινοτόμων στοιχείων έχει ένα κεφάλαιο για την ενέργεια, για τα ενεργειακά θέματα. Αληθεύει ότι η απουσία ενό τέτοιου κειμένου δεν παρακόλλησε στο παρελθόν την ανάπτυξη δευτερογενού νομοθεσία για τα θέματα ενέργεια, βασιζόμενη τότε στι αρμοδιότητε ε, τη ενία εσωτερική αγορά και στο, του περιβάλλοντο, όπω ε, καταδεικνύουν και τα έγγραφα τα οποία διανεμεί θυμήθηκα Αλλά η έναρξη σε ισχύ τη συνθήκη Λισαβόνα μπορεί να σημαίνει μια πολύ σημαντική αλλαγή για τα ενεργειακά θέματα τη Ένωση. Τώρα έχουμε με τη συνθήκη μια νομική βάση που πριν δεν είχαμε <clears throat> και που καθορίζει τα θέματα τα ενεργειακά ω θέματα κοινή ευθύνη στο θέμα αυτό για τον ανεφοδιασμό η συνθήκη της Σαββόνας ε, εισάγει ένα καινοτόμο στοιχείο για την αντιμετώπιση κρίσεων ανεφοδιασμού και με αλληλέγγυο τρόπο να τις ξεπερνάμε. Απ' την άλλη πλευρά η εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενισχύεται με το αξίωμα του του εκπροσώπου <clears throat> καθώς το αναφέρει και η συνθήκη είναι πολύ νωρί σίγουρα για να δούμε πώ αυτό το νέο κείμενο θα επηρεάσει την ενεργειακή πολιτική. Όμω εντωμεταξύ επιτρέψτε μου να αναθεωρήσω και να επισκοπήσω τα θέματα εκείνα τα οποία όσον αφορά την ε, συνθήκη ε, έχουμε ε, σημαντικά στοιχεία μπροστά μα. Τρει πυλώνε θα αναφέρω που θα του αναφέρω ξεχωριστά ενώ όλοι γνωρίζουμε πόσο στενά συνδεδεμένοι είναι αυτοί οι άξονε μεταξύ του. Α γνωρίζουμε επίση από την άλλη πλευρά ότι αυτή η πολιτική θα πρέπει να εξυπηρετεί εξυπηρετεί πάντα τους πολίτες και τους καταναλωτές. Όσον αφορά την, τον, τον ανταγωνισμό, και την αρμοδιότητα για αυτά τα θέματα. Έχουμε ένα πολύ πρόσφατο πακέτο, το τρίτο πακέτο για την εσωτερική αγορά που θα σημαίνει ή σημαίνει ήδη, συνεπάγεται ήδη σημαντικές αλλαγές. Αφενός την διαφοροποίηση με, τρία πρότυπα, με διαφορετικά τρία πρότυπα των υποδομών και της μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας καθώς επίσης και την υπηρεσία συντονισμού των ρυθμιστικών αρχών, ASER. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η προώθηση σε αυτά τα άλλα θέματα <clears throat> έγινε ήδη από την νομοθεσία για τον ανταγωνισμό και την ενιαία εσωτερική αγορά. Χωρίς αμφιβολία ε, η αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι εκείνη που θα ε, ε, παρατηρεί και θα επιτηρεί αυτά τα θέματα. <clears throat> Επίσης έχουν καθοριστεί τα διοικητικά συμβούλια, ο διευθυντής και θα αρχίσει αυτή η υπηρεσία σύντομα να λειτουργεί και παρότι και στην εσωτερική αγορά και στην ε, ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έχουμε συγκεκριμένη νομοθεσία και αυτή σίγουρα συνεισφέρει για την ασφάλεια των εφοδιασμού, σίγουρα αυτή η πτυχή είναι η πιο ευαίσθητη, δηλαδή η ασφάλεια των εφοδιασμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρώτα απ' όλα πρέπει να αναφερθούμε στις ε, υποδομές διασύνδεσης που είναι Θεμελιώδε στοιχείο τη εσωτερική αγορά στην οποία αναφέρθηκα πιο πριν. Σε αυτήν εδώ την περίπτωση τα εθνικά συμφέροντα και τα περιφερειακά συμφέροντα και σε κάποιε περιπτώσει και τα ίδια τα τοπικά συμφέροντα μπορούν να οδηγήσουν σε παράλυση ή να παρακολύσουν την αναγκαία δράση για τα ενεργειακά θέματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέχρι σήμερα βασιζόμαστε με το σημερινό τίτλο 16 για τα ευρωπαϊκά ε, δίκτυα ενέργεια, από πλευρά τη συνθήκη που εντάσσεται στους στόχους ενιαίας εσωτερική αγορά και τη κοινωνική και οικονομική συνοχή. Πέρα από αυτό το όργανο, το μέσο αυτό για τα διευρωπαϊκά δίκτυα, <clears throat> συνεχίζουμε σε πολλέ περιπτώσει να βλέπουμε ότι υπάρχουν δυσκολίε για την διασύνδεση μεταξύ κρατών μελών. Ακριβώ στα σημεία τα κομβικά διασύνδεση, τα διασυνοριακά. Εκεί που είναι πολύ σημαντικό ο χαρακτήρα του. Εδώ πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη αρμοδιότητα από πλευρά των ευρωπαϊκών οργάνων, ώστε να μπορέσει αυτή η κοινή αρμοδιότητα να περάσει στο επίπεδο επίπεδο των Βρυξελών για τη λήψη αποφάσεων. Το βήμα που έγινε τα τελευταία χρόνια με τον διορισμό ε, συντονιστών των προγραμμάτων ήταν ένα σωστό βήμα, <clears throat> αλλά περιορισμένη εμβέλεια. Θα ήθελα να κάνω κάποια σχόλια, συνεχίζοντα την εξέταση αυτού του θέματο. Πρώτα απ' όλα, οι υποδομέ διαδραματίζουν ένα σημαντικό ρόλο στο θέμα του συσχετισμού των σχέσεών μα, των εξωτερικών μα σχέσεων, ιδιαίτερα τη γειτονία και τη συνεργασία. Πρόσφατα στη Μαδρίτη έγινε μια διάσκεψη υψηλού επίπεδου που έγινε, διοργανώθηκε από κοινού από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ισπανική Προεδρία για το θέμα των ενεργειακών υποδομών ως ένα προηγούμενο αναγκαίο βήμα για την πρόταση που ε, εξέφρασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, για, αυτή την, για αυτό το φθινόπωρο για ένα πακέτο υποδομών. <clears throat> Σημαντική διάσταση αυτή. Θεωρούμε ότι μπορεί να χρησιμοποιηθούν επίσης ε, τα μέσα της νέας συνθήκης όσον αφορά την εξωτερική πολιτική ως προς αυτή την κατεύθυνση. Σε σχέση με αυτά χρησιμοποιείται η ρητορία, η διατύπωση να μιλάμε με μία ενιαία φωνή προς το εξωτερικό. Και αυτό θα πρέπει να μεταφράζεται και σε εσωτερικά και εξωτερικά μέσα όπως ε, προβλέπει η δεύτερη αναθεώρηση στρατηγικού χαρακτήρα για τα ενεργειακά θέματα που θα μπορούν να δημιουργήσουν, να κάνουν πραγματικότητα αυτές τις αρχές ε, με ένα συντονισμό και ένα σχεδιασμό που θα είναι αποτελεσματικού χαρακτήρα για τα ενεργειακά θέματα και που θα βασίζονται φυσικά στην πολιτική μας καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών, στην σφαιρική παγκόσμια οικουμενική διάσταση, καθώς επίσης και στα διεθνή φόρα της λέσχης των 20 για παράδειγμα. Χρειάζεται ενιαίες γραμμές, ομοιογενείς γραμμές η Ευρωπαϊκή Ένωση για να είναι αξιόπιστη και να διασφαλίζει την, ε, τις ενεργειακές της ανάγκες. Και αυτό πρέπει να διασφαλίζεται σε ένα ανοιχτό διάλογο με τους κύριους διεθνώς εμπλεκόμενους ώστε οι καταναλωτές και εκείνοι που εφοδιάζουν με ενεργειακά προϊόντα όπως και σε ζώνες διαμετακόμισης να μπορούν να συνεργάζονται. Η ασφάλεια και ο ενεργειακός ανεφοδιασμός θα πρέπει στο μέλλον να αποτελούν ένα θεμελιώδες στοιχείο της εξωτερικής πολιτικής και κοινή ασφάλειας και να είναι αυτά τα μέσα όπως η ε, διπλωματική υπηρεσία ή η υπηρεσία εξωτερικών δράσεων που θα πρέπει να συμμετέχουν. Οι κρίση στον ανεφοδιασμό τα τελευταία χρόνια κατέδειξαν τη σημασία που έχει αυτό το θέμα <clears throat> και που μπορεί να δημιουργούν εντάσεις και τριβές που θα είναι πολύ σημαντικές. Θα ήθελα επίσης να υπενθυμίσω ότι σε αυτόν τον πυλώνα για την ασφάλεια του ανεφοδιασμού βασιζόμαστε ήδη στην παρούσα ενισχύ νομοθεσία καθώς και στην τελική διαπραγμάτευση όσον αφορά τι ε, δράση ε, για τα στρατηγικά θέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου. Επίση, ε, άρχισαν να λειτουργούν οι δράσει σε σχέση με την, το άρθρο τη συνθήκης για το περιβάλλον. Και η ενεργειακή αποτελεσματικότητα και οι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια παίρνουν ένα ιδιαίτερο χαρακτήρα στη νέα συνθήκη. Οι δράσει σε αυτόν τον τομέα γίνονται με βάση πολιτικέ δεσμεύσει στο υψηλότερο, πολιτικό επίπεδο. Το θέμα το οποίο μπορεί να τεθεί εδώ και να εξεταστεί αν η Ευρωπαϊκή Ένωση και πιο συγκεκριμένα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν επαρκείς εξουσίες για να επιτηρούν και να επιβάλλουν τη συμμόρφωση με αυτού του στόχου. Αυτό θα είναι εκείνο το οποίο θα είναι το μήνυμα που θα δώσει στου πολίτε ε, ε, το αίσθημα τη αξιοπιστία και τη ασφάλεια. Δεν μπορούμε να διαχωρίσουμε αυτό το θέμα από τι εξωτερικέ σχέσει που συνδέονται με διεθνεί υποχρεώσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών. Τέλο θα ήθελα να προσθέσω μια τελευταία διάσταση που ίσω όμω είναι πιο σημαντική είναι η διάσταση της τεχνολογίας αυτή. Το έγγραφο του Notre Europe της Ευρώπης μας δείχνει ότι και στην βιομηχανική πολιτική και στην πολιτική τη στρατηγική για την Ευρώπη του 2020 έχουμε μια νέα διάσταση στον τομέα τη ενέργεια. Και ε, χρειάζεται εδώ ένα νέο μέσο από πλευρά τη συνθήκη ε, που έχουμε. Έτσι και σε σχέση με την ανάπτυξη των δράσεων για τη βιομηχανία είναι πολύ σημαντικό το επίπεδο εδώ και σε σχέση με τα ενεργειακά θέματα αυτά τα θέματα αναφέρονται στη χρηματοδότηση περισσότερο σε θέματα χρηματοδότησης. Για τα ενεργειακά θέματα αυτό το πρόγραμμα, αυτό το σχέδιο θα είναι η λιδία λίθο, η μεγάλη δοκιμασία της Ευρωπαϊκής Ένωση. Έχουμε τις ιδέες, τις αναλύσεις και τους προβληματισμούς. Εκείνο το οποίο απομένει να αποφασίσουμε είναι από τους, τομεί ε, από τους τομείς της ιδιωτικής ε, το επίπεδο το οποίο θα αναλάβουν ε, όσον αφορά τις υποχρεώσεις μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, όσον αφορά την ολοκλήρωση τη χρηματοδότηση. Μία ε, θετική ε, είδηση, ένα καλό μαντάτο είναι ότι ε, έγινε στην Μαδρίτη η συνάντηση υπό την Ισπανική Προεδρία την προηγούμενη εβδομάδα με, θετικές, με θετική έκβαση. Κυρίε και κύριοι, εν συντομία έκανα μια επισκόπηση των ενεργειακών θεμάτων σε σχέση με τα μέσα που έχουμε εμεί ω νομοθέτε στη διάθεσή μα. Με τι διατάξει νέα συνθήκη καθώ και με τη δευτερογενή νομοθεσία που πρόσφατα υιοθετήθηκε, πρέπει και μπορούμε να συνεχίσουμε την πορεία μα στα Πραγματικά η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε μια πολιτική πρωτοπορία όσον αφορά την αηφορία με οικονομία χαμηλών εκπομπών ε, άνθρακα και διοξιδίου του άνθρακα λαμβάνοντα υπόψη τον ορίζοντα του 2020 αλλά και πέρα από αυτόν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανήγγειλε το προγραμμα δραση δράσης 2011-2020 κατά τα τέλη ε, του έτου. και θα έχει και την αντίστοιχη ανάλυση και θέματα ελέγχου και επιτήρηση Αξίζει τον κόπο να δούμε με τα ενδιάμεσα αποτελέσματα ώστε όταν θα έρθει η στιγμή να διαπιστώσουμε ποιε είναι εκείνε οι ελλείψει που διαπιστώνονται σε σχέση με τα νομικά μέσα που θα έχουμε στη διάθεσή μας για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις του, του 21ου αιώνα. Θα είναι σίγουρα μια ακρόαση σαν αυτή όπου οι νομοθέτε στο εθνικό επίπεδο και οι ευρωπαϊκοί νομοθέτε συνέρχονται όπου θα πρέπει να εξεταστούν τα θέματα που θα πρέπει να ληφθούν, να αποφασιστούν για το μέλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ουρίμπε. Είστε υπεύθυνο στην κυβέρνησή σας για τα θέματα της ενέργειας, είστε αρμόδιος υπουργός και για την ενέργεια και για τις ιεροδρομικές μεταφορές και τον τουρισμό και αυτά τα οποία είπατε είναι καρπός εμπειρίας θα έλεγα της ε, ισπανικής προοπτικής. Υπάρχουν αρκετά θέματα στην κοινή πολιτική ενέργειας και αυτά που είπατε ήταν ιδιαίτερα χρήσιμα. Μπορείτε να θέσετε εφόσον το επιθυμείτε ε, και ερωτήσεις συνάδελφοι στον εκπρόσωπο του Συμβουλίου. Μετά το τέλος βέβαια ε, των, ε, των ομιλητών. Έχετε τη δυνατότητα μετά να πάρετε το λόγο αρκετοί συνάδελφοι ε, έχουν την δυνατότητα και ορισμένοι το έχουν ήδη ζητήσει να πάρουν το λόγο για τρία λεπτά και μπορούν να καταθέσουν τις ερωτήσεις. Μπορούν και τα υπόλοιπα μέλη ή διάφοροι παρόντες στην αίθουσα να θέσουν ερωτήσεις χρησιμοποιώντας τις ε, ε, μπλε κάρτες. Αλλά για μια ακόμη φορά έχω την τιμή να σας παρουσιάσω τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Χωακίνα Μόλια ο Χακίν Αλμούνια εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον τομέα του ανταγωνισμού. Πώς μπορούν να βελτιωθούν οι συνθήκες του ανταγωνισμού. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να υπάρξουν ξεκάθαροι κανόνες, απλοί κανόνες για τη λειτουργία της αγοράς. Αυτό έχει σημασία για τις εταιρείε που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ενέργειας, για τις μικρότερες εταιρείε, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και για τον ίδιο τον πολίτη απαιτείται να υπάρχει ελεύθερος ανταγωνισμός έτσι ώστε να μειώσουμε το κόστος της ενέργειας. Η ανταγωνιστικότητα βέβαια είναι πάρα πολύ περίπλοκο πράγμα και θα θέλαμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνει συνολικά ανταγωνιστική. Κύριε Αντιπρόεδρε λοιπόν, περιμένουμε με πολύ ενδιαφέρον τις παρατηρήσεις σας. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την Ισπανική Προεδρία και όλους εσάς επίσης που με προσκαλέσατε να συμμετάσχω. Πολύ περίπλοκο είναι. Συγγνώμη, αυτό το κουμπί εδώ, αυτό το μικρόφωνο. εντάξει, ζητώ συγγνώμη. Επαναλαμβάνω, Πρόεδρε. <clears throat> Πρόεδρε, σα ευχαριστώ πολύ για αυτή την πρόσκληση να συμμετάσχω από κοινού με την Ισπανική Προεδρία και τα Εθνικά Κοινοβούλια και το ίδιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε αυτό το ημικύκλιο, σε αυτή την αίθουσα τη Ολομέλεια, σε μια ανταλλαγή απόψεων, ιδεών, προτάσεων, κατευθυντηρίων γραμμών για κάτι που είναι τόσο σημαντικό για όλου εμά ω ε, ε, Ευρωπαίοι που είμαστε, όπω είναι η ευρωπαϊκή πολιτική στα ενεργειακά θέματα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζουμε απόλυτα και πλήρω το όραμα και την προσέγγιση μια ευρωπαϊκή πολιτική στα ενεργειακά θέματα που θα βασίζεται σε τρει πυλώνε, σε τρει ουσιώδει άξονε για τους οποίους έγινε ήδη λόγος από τους εισηγητές ε, ε, των ομάδων ε, των κύκλων εργασιών και από τον εκπρόσωπο της Προεδρίας του Συμβουλίου. Πρώτα απ' όλα την ασφάλεια στον ανεφοδιασμό στα ενεργειακά θέματα που έχει ρόλο κλειδιού. Και είναι σαφέ και είχαμε ευκαιρία σε πραγματικό χρόνο να διαπιστώσουμε τα προβλήματα τα οποία ετίθενται στους ε, έναντι των Ευρωπαίων πολιτών για εκατομμύρια Ευρωπαίους πολίτες προβλήματα υπερβολικής εξάρτησης όσον αφορά ενεργειακά προϊόντα από το εξωτερικό που δημιουργούσαν ανασφάλεια σε σχέση με τον πρωτογενή ανεφοδιασμό με φυσικό αέριο τη της ε, Ευρώπης στα προηγούμενα χρόνια. Δεύτερος ουσιώδης πυλώνας, η ανταγωνιστικότητα, ο ανταγωνισμός. Είναι αυτονόητο αυτό. Και τρίτον, επίση, αλλά εξίσου σημαντικό, τελευταίο, αλλά εξίσου σημαντικό η αηφορία. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, χάρη στι πρωτοβουλίε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και χάρη στι συζητήσει σε βάθο που έγιναν για τα θέματα που συνδέονται με την αηφορία, και έγιναν εδώ στην Ευρωβουλή και στο Συμβούλιο αυτέ οι συζητήσει, η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν χάρη σε αυτές τις πρωτοβουλίε ικανή να βρει μια σύνθεση και μια σύγκληση κατεύθυνσης ισχυρή μεταξύ των ενεργειακών αναγκών των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, των νέων τεχνολογιών για τα θέματα τα ενεργειακά και από την άλλη πλευρά την αηφορία όσον αφορά το περιβάλλον και ιδιαίτερα την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών. Και πιστεύω ότι αυτό μας έκανε εμάς όχι μόνο ένα χώρο, δημιούργησε από την Ευρώπη ένα χώρο όπου οι δύο αυτοί οι στόχοι συντονίζονται επαρκώς με στόχους και μέσα για την επίτευξή τους, αλλά είμαστε και πρωτοπόροι και ηγέτες σε παγκόσμια κλίμακα. Σε αυτή τη μάχη που δίνουμε να συγκλίνουν οι στόχοι των ενεργειακών πόρων και της καταπολέμησης των κλιματικών αλλαγών και του σεβασμού του περιβάλλοντος. Έτσι, με αυτούς τους ε, πυλώνες η ενέργεια πρέπει να έχει προσιτές τιμές, να είναι προσιτή για όλους. Και σε αυτό το σημείο διαδραματίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο χωρίς αμφιβολία η πολιτική για τον ανταγωνισμό <clears throat> για την οποία είμαι αρμόδιος ε, άμεσα επίτροπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά <clears throat> σε αυτή την αρχική παρέμβαση θα τοποθετηθώ γενικότερα στην ενεργειακή πολιτική και όχι υπό το στενό πρίσμα του ανταγωνισμού υπό το πρίσμα του προγράμματος εργασίας που έχει υποβάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και που έχει συζητηθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν από κάποιους λίγους μήνες σε σχέση με τη νέα Επιτροπή που ξεκίνησε να λειτουργεί <coughs> στις 10 Φεβρουαρίου εφέτος. Λάβαμε λοιπόν υπόψη αυτές τις αρχές εμείς και ταυτόχρονα επίσης τους εντάξαμε αυτούς τους στόχους στην πρότασή μας για μια ευρωπαϊκή στρατηγική ανάπτυξης αποτελεσματικής ανάπτυξης, ανταγωνιστικής δυναμικής ανάπτυξης με κοινωνική ένταξη και ολοκλήρωση και συνεκτική και σε συνοχή με τους στόχους σεβασμού του περιβάλλοντος και της προστασίας του. Αυτή είναι η στρατηγική για την Ευρώπη του 2020 που την επόμενη εβδομάδα ελπίζω ότι τελικά θα εγκριθεί και θα υποστηριχθεί από το <clears throat> Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τους 27 αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δράσαμε λοιπόν τους τελευταίους χρόνους με έντονους ρυθμούς ε, για να προχωρήσουμε σε μια ευρωπαϊκή πολιτική για τα ενεργειακά θέματα. Αλλά έχουμε συνειδητοποιήσει και γνωρίζουμε ότι αυτή οι έντονοι ρυθμοί πρέπει να διπλασιαστούν και πάλι εν ώψη των μελλοντικών προκλήσεων. Εργαζόμαστε για την ανάπτυξη μια στρατηγική εξειδικευμένη, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Και θα συγκεκριμενοποιήσουμε αυτή τη στρατηγική μα ιδιαίτερα στο πρόγραμμα δράσεω για τα ενεργειακά θέματα, στο οποίο μόλι ε, έκανε αναφορά ο Πέντρο Μαρίν πιο πριν. Στο πρόγραμμα δράση λοιπόν για την ενεργειακή αποδοτικότητα και τον οδικό μας χάρτη <clears throat> μακροπρόθεσμα πώς πρέπει να κινηθούμε για να πετύχουμε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα το 2050 σε, ε, που να συνάδει με τους, ε, τις παγκόσμιες υποχρεώσεις, τις υποχρεώσεις που έχουμε επομιστεί σε παγκόσμια κλίμακα. Αυτό το σύνολο μέτρων λοιπόν θα μας εξυπηρετήσει, πρέπει να εξυπηρετήσει για να ταυτοποιήσουμε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα επόμενα χρόνια τις προκλήσεις του μέλλοντος. Όμως, το γεγονός ότι θα έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας, αυτό δεν σημαίνει από την άλλη πλευρά ότι δεν καταφέραμε εμείς τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να δουλέψουμε και να δράσουμε μέσα στο νομικό πλαίσιο που ισχύει σήμερα αποτελεσματικά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πριν αρχίσει να ισχύει η συνθήκη της Λισαβόνας ήδη είχε σημαντικές βάσεις, σημαντικές για να δραστηριοποιηθεί. Και τώρα, όπως είπαν και οι συγητές, και ο Υφυπουργό από την Ισπανική κυβέρνηση, από την Ισπανική Προεδρία, έχουμε μια νέα νομική βάση για την ενέργεια πλέον, για τα ενεργειακά θέματα, που ισχύει από τότε που άρχισε να ισχύει η συνθήκη της Λισαβόνα, την 1η Δεκεμβρίου το 2009. Όμω θα ήθελα να εμείνω και να επιμείνω στο γεγονό ότι πριν ακόμα αρχίσει να ισχύει η συνθήκη τη Λισαβόνα, πριν αρχίσει να ισχύει, η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν ικανή να αναπτύξει μια ενεργειακή πολιτική στεναρή και αποτελεσματική με, τη βάση, με βάση τριών αρχών, θεμελιωδών αρχών, στι οποίε αναφερθήκαμε πιο πριν. Και δρώντα ταυτόχρονα όχι μόνο για τα θέματα ανταγωνιστικότητα και ανταγωνισμού, για την ασφάλεια του ανεφοδιασμού και την αηφορία, αλλά επίση ε, εγγυόμενοι και προσπαθώντας να εγγυηθούμε στο μέτρο των δυνατοτήτων και ικανοτήτων μας προσιτές τιμές για τα ενεργειακά προϊόντα και την χρήση τους και για τους καταναλωτές και ταυτόχρονα για τους χρήστες ενεργειακών πόρων στο παραγωγικό μας βιομηχανικό σύστημα. Υπό αυτό το πρίσμα είναι πολύ σκόπιμο και σημαντικό να αναφερθώ στο τρίτο νομοθετικό πακέτο για την, για αγορά φυσικού αερίου και ενεργειακών πόρων που εγκρίθηκε κατά την τελευταία φάση της προηγούμενης ε, εντολής. Η υλοποίηση των μέτρων αυτών τώρα ε, γίνεται και από τα εθνικά κοινοβούλια και από τις ε, εθνικές αρχές. Αυτή η μεταφορά στο εθνικό επίπεδο θα ολοκληρωθεί, πρέπει να, ολοκληρωθεί πριν από το Μάρτιο 2011. Έχουμε 19 μήνες ακόμα για να ολοκληρώσουμε την ε, υλοποίηση του τρίτου νομοθετικού πακέτου στα 27 κράτη-μέλη. Και εμείς θεωρούμε υπό το δικό μας πρίσμα αυτή, αυτός θα είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της ενεργειακής πολιτικής που θα πρέπει να βασίζεται σε μια ορθή μεταφορά και μετάθεση έγκαιρα και το δυνατόν πιο φιλόδοξη αυτών των μέτρων αυτού του πακέτου. Ταυτόχρονα παράλληλα με αυτό αναπτύσσουμε και σε ευρωπαϊκή κλίμακα αλλά και σε σχέση με συζητήσεις και τις διαβουλεύσεις που έχουμε με του εταίρους μα σε παγκόσμια κλίμακα το πακέτο μέτρων για την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών και τα ενεργειακά θέματα. Έχουμε το πακέτο 2020-2020, ε, έχουμε την αναθεωρημένη οδηγία σε σχέση με την ε, ενεργειακή εκμετάλλευση κτηρίων, έχουμε την οδηγία για την ε, αποτελεσματικότητα στην τελική χρήση ενέργειας και ενεργειακών πόρων, όλα αυτά μέσα σημαντικά και θεμελιώδη που ήδη εγκρίθηκαν και έχουν εγκριθεί. Και αυτό που πρέπει τώρα να γίνει είναι να μεταφερθούν στις εθνικές νομοθεσίες και να λειτουργήσουν εκεί όπου πρέπει. Και κυρίως η εφαρμογή τους είναι σημαντικό στοιχείο. Εξίσου ταυτόχρονα είναι αναγκαίο να αναπτύξουμε στο σύνολο την, ε, μια οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ένα θέμα τεράστιας σημασίας, <clears throat> χωρίς το οποίο δεν θα μπορέσουμε να πετύχουμε τους στόχους που έχουν καθοριστεί για το 2020. Επιπλέον, παράλληλα με όλα αυτά, έχουμε τη νέα νομική βάση της συνθήκης. Αναφέρθηκε αυτό. Το άρθρο ιδιαίτερα 194 της συνθήκης στο οποίο πρέπει να προσθέσουμε την ρητή αναγνώριση για την αρμοδιότητα, νομική αρμοδιότητα από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης σε περίπτωση κρίσης για θέματα ενεργειακών ανεφόδιασμού που, αναφέρεται στο άρθρο της ε, ε, συνθήκης της Λισαβόνας ε, και όπως το γνωρίζουμε σήμερα εμείς. Και γι' αυτό λοιπόν έχουμε μέσα και μέτρα που μπορούν να λειτουργήσουν μέσα στο πλαίσιο μιας στεναρής ε, αποτελεσματικής πολιτικής και που πρέπει να υλοποιηθούν. Έχουμε νέες νομικές βάσεις. Αυτό που πρέπει τώρα να γίνει είναι να γίνει κάθε προσπάθεια από πλευρά μας να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Αυτό σημαίνει σε πολλές περιπτώσεις να είμαστε πιο συντονισμένοι σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε μεγαλύτερο βαθμό να υπάρξει συντονισμό για την επίτευξη αυτών των στόχων. Αυτών των στόχων που εδώ εγκρίθηκαν στα εθνικά κοινοβούλια και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο όλο αυτό το σύνολο των μέτρων να υλοποιηθεί. Επιμένω και μένω για τη σημασία που έχει να μπορέσουμε το Μάρτιο του 2011 να καταλήξουμε σε ένα βαθμό το οποίο θα είναι ο υψηλότερος δυνατός στην ε, υλοποίηση των μέτρων του πακέτου. Με όλα αυτά θα βοηθήσουμε θα βοηθήσουμε να εμβαθύνουμε στην ενιαία εσωτερική αγορά ενεργειακών θεμάτων. Να εμβαθυνθεί αυτή η αγορά. Είναι ένα στόχο κλειδί αυτό. Η έκθεση Μόντι που πρόσφατα παρουσιάστηκε πριν από κάποιε λίγε εβδομάδε και που σημαίνει μια νέα ανάγνωση των φιλοδοξιών και των προσδοκιών που πρέπει να έχουμε ως Ευρωπαίοι για να έχουμε μια πραγματική αυθεντική ενιαία εσωτερική αγορά με 500 εκατομμύρια πολιτών που θα είναι χρήστες, καταναλωτές, οικονομικά εμπλεκόμενοι σε αυτή την έκθεση Μόντι αναφέρονται τα θέματα των φραγμών και εμποδίων. Αναφέρονται τα θέματα που εκκρεμούν. Αναφέρονται οι δυνατότητες για την υπέρβαση και επίλυση αυτών των προσκομμάτων και των ε, εμποδίων και φραγμών. Και πολλοί που το προανέφεραν υπάρχουν θέματα που εκκρεμούν για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια ενιαία εσωτερική αγορά ενεργειακών πόρων. Ιδιαίτερα υπάρχουν θέματα που εκκρεμούν και είναι πιο κατεπίγοντα όσον αφορά την ε, ε, απουσία διασύνδεσης ε, μεταξύ ζωνών και περιφερειών μέσα στην ίδια την ευρωπαϊκή επικράτεια και υπό το ιδιαίτερο πρίσμα αυτό υπάρχουν προσκόμματα και φραγμοί όσον αφορά την απουσία ανταγωνισμού όπου ακόμα δεν υπάρχει η πλήρης χρήση και λειτουργία των κανόνων του ανταγωνισμού όσον αφορά τα παλαιότερα μονοπόλια ή κονσόρτσια ή κρατικά μονοπόλια που δεν χρησιμοποιούν όπως θα έπρεπε σύμφωνα με τις διατάξεις και τις συνθήκες της ε, συστράσεις τους τα θέματα των επιδοτήσεων και κρατικών ενισχύσεων όσον αφορά την μεταφορά ή ε, ε, διανομή μέσα από το δίκτυο των, ε, της ηλεκτρικής ενέργειας. Αλλά η ενιαία εσωτερική αγορά δεν θα γίνει εν μια νυχτή, το γνωρίζουμε αυτό λόγω της πείρας μας. Και υπάρχει ένας τρόπος να προχωρήσουμε προς την ενιαία εσωτερική αγορά ενέργειας, στον οποίο τρόπο και μέσω δίνουμε την αναγκαία προσοχή από πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό ο τρόπο είναι η περιφερειακή συνεργασία. Η περιφερειακή συνεργασία είναι σκόπιμη και είναι αποτελεσματική σε συγκεκριμένε περιφέρειε και περιοχέ των κρατών μελών μεταξύ συγκεκριμένων κατηγοριών των κρατών μελών. Είναι δυνατόν μέσα στο πλαίσιο των να υπάρξει αυτή η περιφερειακή συνεργασία και είμαστε πεισμένοι ότι πέρα από τα άμεσα ωφέλη για όσους θα συμμετέχουν άμεσα σε αυτή την περιφερειακή συνεργασία στα ενεργειακά θέματα αυτή η οδός είναι μια ένα σημαντικός μοχλός που δίνει αποτέλεσμα μοχλικό μόχλευσης και δίνει δυνατότητα επίτευξης μεγαλύτερου ρυθμού και μεγαλύτερης ταχύτητας και αποτελεσματικότητας όσον αφορά την επίτευξη της ενιαίας εσωτερικής αγοράς. Είναι αυτονόητο ότι μια ενιαία εσωτερική αγορά όσον αφορά τα ενεργειακά θέματα για να λειτουργεί σωστά θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την εξωτερική διάσταση. Αφενός κάνοντα χρήση τη ε, διάσταση ε, αυτή για να επιληθούν καλύτερα τα θέματα ε, ανεφοδιασμού μας στον πρωτογενή τομέα με ενεργειακά προϊόντα από το εξωτερικό και κατά δεύτερο λόγο για να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα, το δυναμικό των κρατών μελών στις σχέσεις τους με εξωτερικές αγορές υπό ε, πολυσχηδές πρίσμα αυτό με πολύμορφο τρόπο. Εργάζεται έντονα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να εξευρωπαίσει τα συμφέροντα των κρατών μελών στις σχέσεις τους με το εξωτερικό όσον αφορά θέματα ανεφοδιασμού αλλά όσον αφορά και θέματα αγορών επίσης και πιστεύουμε και θεωρούμε ότι το νέο θεσμικό μέσο, η νέα αυτή θεσμική δυνατότητα που παρέχει η συνθήκη της, της Λισαβόνας και ιδιαίτερα η παρουσία και ύπαρξη του ύπα του εκπροσώπου που παράλληλα με την ιδιότητα του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θα έχει δίνει την δυνατότητα να είμαστε πιο αποτελεσματικοί σε ένα στοιχείο που έχει σημασία κλειδιού και που περιγράφεται σαφώς στον πρόλογο που συνέταξε ο Ζακ Ντελόρ για την έκθεση Notre Europe που παρουσιάστηκε χθε εδώ σε αυτή την συνεδρίαση. Ολοκληρώνω Πρόεδρε. Ολοκλήρωσα. Και πάλι ευχαριστώ πολύ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που διοργάνωσε αυτή τη συνεδρίαση. Συνεδρίαση και που μα προσκάλεσε εδώ σήμερα και χθε. Ευχαριστώ πολύ του εκπροσώπου των Εθνικών Κοινοβουλίων που προσήλθαν σε αυτόν τον διάλογο χάρη στην Ισπανική Προεδρία του Συμβουλίου <clears throat> με τη συνθήκη τη Λισαβόνα που άρχισε να λειτουργεί αυτό ο διάλογο μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Εθνικών Κοινοβουλίων και πέρα από το Κοινοβούλιο, μεταξύ των θεσμικών οργάνων κιόλα τη Ευρωπαϊκή Ένωση ε, σε κοινοτική κλίμακα και των εθνικών κοινοβουλίων αυτό ο διαρθρωμένο διάλογο είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να είναι η εξαίρεση αλλά ο κανόνα. Και όχι μόνο επειδή όπω στα θέματα τα ενεργειακά έχουμε πολλέ κοινέ αρμοδιότητε, συμμεριζόμενε αρμοδιότητε, αλλά και επειδή ο διάλογο των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων και των ε, Ευρωπαϊκών Κοινοβουλίων ε, είναι ένα μέρο τη λύση, όχι όλη το σύνολο τη λύση, αλλά ένα μέρο τη επίλυση των προβλημάτων στο να περάσει προ του πολίτε το μήνυμα που πρέπει να του δώσουμε. Το για το τι σημαίνει η Ευρώπη, τι είναι αυτό που είναι η Ευρώπη και τι κάνει και ποιοι είναι οι στόχοι τη και πώ μπορεί να συνεισφέρει η Ευρώπη για να βελτιωθεί η ζωή των πολιτών στο μέλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να μου επιτρέψετε να σας θυμίσω ότι μπορείτε να ζητήσετε το λόγο, προβλέπετε. Υπάρχουν τα ειδικά χαρτάκια τα οποία μπορεί να θέσουν στη διάθεσή σας οι εκπρόσωποι της γραμματείας. Εφόσον λοιπόν έχετε κάποιες συγκεκριμένες ε, ερωτήσεις να κάνετε προς τους ομιλητές, μπορείτε να σηκώσετε την μπλε κάρτα σας. Θα ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Θυμίζω εδώ ότι ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου και ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι παρόντες και θα δεχθούν τις ερωτήσεις σας. Ο κύριος, ο εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει το λόγο. Ο κύριος Μπαλτσίτης. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, συνάδελφοι από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από τα Κοινοβούλια των κρατών μελών. Θα ήθελα ξεκινώντας να σας ευχαριστήσω για την πρωτοβουλία την οποία πήρατε, για την συνάντηση αυτή την οποία κρίνω ιδιαίτερα επίκαιρη. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ισπανική Προεδρία αναγνωρίζουν την ύπαρξη των προβλημάτων και ε, πράγματι οι συγητές από τις τρεις ομάδες εργασίας μας παρουσίασαν απόψεις τις οποίες θα χαρακτήριζα κυρίως επαγγελματικού επίπεδου θα έλεγα. Η εμπειρογνωμοσύνη τους είναι εντυπωσιακή. Τα προβλήματα είναι γνωστά. Υπάρχει μια, θα έλεγα σε ορισμένες περιπτώσεις, ενεργειακή απομόνωση περιοχών. Υπάρχει ένα πρόβλημα σχετικά με την διασφάλιση της προμήθειας ενέργειας. Υπάρχουν προβλήματα με την τιμολόγηση της ενέργειας και πάει λέγοντας. Υπάρχουν πολλά ακόμα χαίνοντα προβλήματα στον τομέα της ενέργειας. Το θέμα της δικτύωσης των δικτύων ενέργειας είναι ένα θέμα πάρα πολύ περίπλοκο. Οι επενδύσεις στον τομέα αυτό είναι επενδύσεις οι οποίες είναι ιδιαίτερα υψηλού κόστους. Υπάρχει θα έλεγα και μια έλλειψη σχετική πολιτικής βούλησης και όλα αυτά είναι μόνιμα εμπόδια στο να υπάρξει μια πραγματική κοινοτική αντιμετώπιση. Οι νέες τεχνολογίες, η πράσινη τεχνολογία είναι θέματα στα οποία θα πρέπει να ενσκύψουμε στο μέλλον, αντιμετωπίζοντας όμως πρώτα το θέμα της έλλειψης πολιτικής βούλησης. Το τρίτο πακέτο για την ενέργεια είναι πολύ φιλόδοξο βέβαια και αν εφαρμοστούν οι προτάσεις οι οποίες περιλαμβάνονται τότε θα μπορέσουμε να λύσουμε αρκετά από τα πιο απλά τουλάχιστον προβλήματα. Εάν δεν υπάρξει μια κυρίαρχη εσωτερική αγορά στην ενέργεια, θα χάσουμε πόντους στο επίπεδο του ανταγωνισμού σαφέστατα. Πρέπει να δημιουργηθεί η ενιαία αγορά της ενέργειας, πρέπει να ξεκινήσουμε με συγκεκριμένα βήματα, μικρά βήματα, σαν παράδειγμα αγορές ποσοτήτων φυσικού αερίου όταν συζητάμε τα θέματα της προμήθειας φυσικού αερίου με εξωτερικούς προμηθευτές. Μπορούμε να συνδυάσουμε τα συμφέροντα των κρατών μελών. Θα πρέπει επίσης τα θέματα της ενέργειας στο μέλλον όταν τα συζητάμε να τα συνδέουμε με την δυνατότητα παρέμβασης την περίπτωση όπου δημιουργούνται φυσικές καταστροφές όπως αυτές, σαν παράδειγμα που γνωρίζουμε τον τελευταίο καιρό στον κόλπο του Μεξικού. Αν υπήρχε μια συνεργασία κρατών στην περιοχή, η απάντηση μπορεί να ήταν πιο αποτελεσματική. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Μπαλτσούτης. Ο επόμενος εκπρόσωπος προέρχεται από την Τουρκική Βουλή, ο κύριος Κυράν. Η ενέργεια είναι ένα βασικό συστατικό, θα έλεγα, όλων των οικονομικών τομέων. Είναι κάτι το οποίο επηρεάζει άμεσα την καθημερινότητά μας. Δεν μπορούμε εμείς να προχωρήσουμε στην κοινωνική και οικονομική πρόοδο αν δεν έχουμε διασφαλίσει τα προβλήματα της ενέργειας. Για την αηφόρο επίσης ανάπτυξη η διασφάλιση της προμήθειας ενέργειας είναι βασικό ε, συστατικό. Θα πρέπει να υπάρξει και διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας όπως και διαφοροποίηση των προμηθευτών. Το κόστος της ενέργειας και η ασφάλεια στον τομέα της ενέργειας εξαρτάται κυρίως ε, από την ε, ένταση που χαρακτηρίζει την αγορά ενέργειας και από την ασφάλεια επίσης που την χαρακτηρίζει. Ο προγραμματισμός των μελλοντικών αναγκών μας σε ενέργεια ε, θα πρέπει να λάβει υπόψη ότι οι υδρογονάνθρακες οι οποίοι είναι διαθέσιμοι ε, δεν ε, είναι κάτι το οποίο απεριόριστα θα ανανεούται. Ας πούμε ότι έχουμε την δυνατότητα χρήσης υγρών καυσίμων για τα επόμενα 40 χρόνια και αερίου για τα επόμενα 60 χρόνια. Η αποτελεσματικότητα της ενέργειας και σε επίπεδο παραγωγής και σε επίπεδο χρήσης πρέπει να είναι βασικό χαρακτηριστικό της πολιτικής μας. Σαν μελλοντικός εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Θα έλεγα ότι αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η προστασία του περιβάλλοντος, η οργάνωση της εσωτερικής αγοράς και η καλύτερη διαδικτύωση. Αλλά όλα αυτά είναι αρκετά, αναρωτιέμαι για να μπορέσει η ευρωπαϊκή κοινότητα ενέργειας η οποία ξεκινάει να σταθεί αποτελεσματικά. Είναι απαραίτητο να συνεργαστούν και τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Και αυτές οι χώρες θα πρέπει για να μπορέσουν να συνεργαστούν με την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, να έχουν κοινά σύνορα με την Ένωση. Οι υποψήφιες χώρες. Ξέρετε ότι εμείς είμαστε σε τελωνιακή ένωση με την Ευρωπαϊκή Ένωση από το 1995. Θα προσκληθούμε Ξέρετε επίσης πως η σημασία των κοιτασμάτων φυσικού αερίου του Ιράν και του Ιράκ είναι κεφαλαιόδους σημασίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορούμε λοιπόν και σαν Τουρκία να παίξουμε έναν ρόλο έτσι ώστε να εξομαλύνουμε τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες αυτές και να βοηθήσουμε και τον εκδημοκρατισμό των χωρών αυτών. Να μην ξεχνάμε επίσης και τον αγωγό Ναμπούκο. Ε, δεν συνδέω με το θέμα του Ναμπούκο με τις διαπραγματεύσεις ε, με τις ενταξιακές. Τελειώνω κύριε Πρόεδρε. Αλλά όλα αυτά δεν μπορεί να αγνοηθούν όταν ληφθούν οι τελικές αποφάσεις. δεν καταλαβαίνουμε γιατί εδώ και αρκετό καιρό δεν ανοίγει το κεφάλαιο για την ενέργεια ενώ δεν υπάρχουν τεχνικά εμπόδια γύρω από αυτό. Παρακαλώ να είστε πιο σύντομοι. Ο συνάδελφος από τη Βουλή των Ελλήνων έχει το λόγο για να θέσει την ερώτησή του. Έχετε 30 δευτερόλεπτα. Ήθελα να κάνω μια ερώτηση στον εκπρόσωπο του Συμβουλίου. Κατά πόσο πιστεύει ότι η μακροπρόθεσμα η απελευθέρωση της ε, αγοράς ηλεκτρισμού θα συμβάλλει στην πτώση των τιμών. Και αυτό το λέω ε, επειδή ε, δαιμονοποιείται ο άνθρακας και θα αυξηθεί το κόστος ενέργειας από τις ανθρακικές μονάδες λόγω επιβολής προστήμων διοξιδίου του άνθρακα ε, από την άλλη πλευρά τα υγρά καύσιμα και το αέριο ανεβαίνουν οι τιμές και η διείσδυση στο σύστημα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα είχε ως αποτέλεσμα την άνοδο της τιμής. Κατά πόσο λοιπόν είναι αισιόδοξο ότι ο ανταγωνισμός θα συμβάλλει στη μείωση της τιμής στον καταναλωτή και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την ερώτησή σας αγαπητοί συνάδελφοι αν έχετε γενική ερώτηση και όχι σε σχέση με έναν συγκεκριμένο ομιλητή δηλαδή τον ομιλητή που μόλις παρενέβη παρακαλώ να μην είναι ερωτήσεις για το τέλος διότι αυτή η ερώτηση δεν είχε άμεση σχέση με την ε, ερώτηση σχετικά ε, με ε, τον συνάδελφο από την Τουρκία. Οπότε, εάν αναφέρεστε ε, σε σε ένα συγκεκριμένο θέμα ε, σηκώστε την μπλε κάρτα σας. Αν έχετε γενική ερώτηση όμως σαν αυτήν, παρακαλώ να περιμένετε στο τέλος. Όλοι θα έχουν χρόνο για να απαντήσουν και επίσης ε, για να υπάρχουν ερωταπαντήσεις γενικώ. Ο επόμενος ομιλητής, εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, συνάδελφος Ορέστε Ρώση, έχει το λόγο. Αγαπητοί συνάδελφοι, τελειώνει σχεδόν η συνάντησή μας για την ενέργεια. Ελπίζω να ήταν χρήσιμη έτσι ώστε να ανοίξουν επαφές ανάμεσα στα Εθνικά Κοινοβούλια και τα Κοινοβούλια, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Από τη θέση ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας τα πράγματα έχουν αλλάξει και για τις χώρες μας και είμαστε υποχρεωμένοι να προχωρήσουμε σε στενό διάλογο. Non Ας μην ξεχνάμε λοιπόν ότι η ενέργεια και το περιβάλλον συνδέονται πάρα πολύ στενά, όπως συνδέονται επίσης και με την οικονομία. Δεν θα πρέπει λοιπόν να επιμένουμε σε ιδιαίτερα ακριβές παρεμβάσεις οι οποίες δεν οδηγούν σε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Στην Επιτροπή Περιβάλλοντος συζητάμε τον κανονισμό για τις εκπομπές καυσαερίων από τα ελαφρά εμπορικά οχήματα για να μπορέσουμε να μειώσουμε κατά 5 τουλάχιστον τις 100 στα επόμενα χρόνια τις εκπομπές αυτές. Αν ο κανονισμός γίνει δεκτός όπως προτείνεται θα επηρεάσει αρνητικά την βιομηχανία αυτοκινήτων και θα προκαλέσει μια ζημιά 45 δισεκατομμυρίων ευρώ λέει ο μιλητής. Καταλαβαίνετε ότι ένα τέτοιο κόστος, η μείωση την οποία θα έχουμε πετύχει σε παγκόσμιο επίπεδο, ακούστε, θα είναι περίπου κατά 0,0014%. Αυτό θα έχουμε κερδίσει, δηλαδή τίποτα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλες οι ανθρώπινες δραστηριότητες σε παγκόσμιο επίπεδο δεν αντιπροσωπεύουν πάνω από το 4% της εκπομπής καυσαερίων. Είναι λοιπόν καλύτερο να χρησιμοποιούμε τα χρήματα που έχουμε στη διάθεσή μας για σωστότερους στόχους, νέες τεχνολογίες, νέες μορφές ενέργειας, νέες μονάδες παραγωγής με χαμηλή ενεργειακή ανάγκη και να ευνοήσουμε την έρευνα, να χρηματοδοτήσουμε την έρευνα. Η έρευνα θα μας βοηθήσει να ξεφύγουμε από τα προβλήματα. Η κυρία Μέρκελ, ξέρετε, έκανε προτάσεις δημοσιονομικές. Σε όλους τους τομείς προβλέπονται μειώσεις για τα επόμενα χρόνια, εκτός από την έρευνα. Και ε, το 2009, την ε, χρονιά της μεγάλης κρίσης στις Ηνωμένε Πολιτείες, Όλα ε, υπέστησαν μειώσεις στις Ηνωμένε Πολιτείε από πλευρά της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης, εκτός από την έρευνα. Η έρευνα έφτασε σε δυσθεώρητα ύψη η χρηματοδότησή της. Λοιπόν, κλείνω εδώ. Θα ήθελα να αναφερθώ ιδιαίτερα στην ε, παρουσίαση των εργασιών της Ομάδας Εργασίας Υπαριθμού 3. Υπάρχει θέμα με την ανταγωνιστικότητα και με την αηφορία και με την διασφάλιση φυσικά των προμήθειας ενέργειας. Αυτές οι τρεις ε, βάσεις θα έλεγα είναι οι παράγοντες που θα χαρακτηρίσουν την ενέργεια στην Ευρώπη. Αν δεν λύσουμε τα προβλήματα που υπάρχουν σε αυτούς τους τρεις τομείς τότε δεν θα είμαστε ισχυροί στην παγκόσμια αγορά. και νομίζω ότι οικονομικά αυτό θα προκαλέσει προβλήματα όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και στις φίλες χώρες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την δήλωσή σας και τώρα ο κύριος Έντσελ και πάλι από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εισηγητές για τις εκθέσεις τους και τον Υφυπουργό Ουρίβα και τον Επίτροπο Αλμούνια για τις παρουσιάσεις τους διότι αντιλαμβάνομαι ότι στηρίζουν το εγχείρημά μας και ε, όταν εσείς κύριε πρόεδρε Μπούζε ξεκινήσατε αυτή τη διαδικασία όταν μας το αναφέρατε πριν από μερικές εβδομάδες στο Στρασβούργο ήμουν πολύ απεσιόδοξος για την υλοποίηση αυτής της ενεργειακής ευρωπαϊκής κοινότητος αλλά πιστεύω ότι πολλά ερωτήματα έχουν εντωμεταξύ απαντηθεί μέχρι σήμερα και το πρόγραμμα αυτό είναι εφικτό και είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο θα μπορέσουμε να επιλύσουμε το ενεργειακό ε, για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το οποίο με απασχολεί σήμερα είναι κάτι αρκετά σημαντικό, δηλαδή η κοινωνική πτυχή την οποία δεν πρέπει να ξεχνάμε, πρέπει να την έχουμε στο νου μας στην ε, νέα αυτή ε, δραστηριότητα διότι υποθέτω ότι θα ληφθούν μέτρα, θα υπάρχει απελευθέρωση των αγορών η οποία θα οδηγήσει σε ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο. Θα πρέπει να ρυθμιστούν οι τιμές σε τομείς όπου η αγορά δεν μπορεί να καλύψει κοινωνικώς αποδεκτά τα όρια των κρίσεων και θα πρέπει ίσως να υπησέλθουν και οι ιδιώτες επενδυτές ε, για την ενίσχυση Τη της υποδομής. Ε, θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση και των εμπλεκομένων και των Ευρωπαίων πολιτών. Το ερώτημα είναι αν οι οργανώσεις αυτές, οι εταιρείε αυτές ε, θα ε, είναι αλληλέγγυοι με τους καταναλωτές τους οποίους απευθύνονται και με τα κράτη-μέλη όπου εξασκούν τις δραστηριότητες τους. Οι εταιρείε αυτές θα μπορέσουν να δεχτούν κάποια εποπτεία ε, από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα διότι δεν θα μπορέσουν να υπάρξουν εξαιρέσει εάν μία εταιρεία ε, αρνηθεί τον έλεγχο θα είναι ε, persona non grata δεν θα είναι ευπρόσδεκτη και θα πρέπει οι εταιρείε να το αντιληφθούν και ε, να ε, μπορέσουν ε, να λάβουν υπόψη την κοινωνία και να τις αποδώσουν όσα έχουν λάβει από αυτήν. Και όταν μιλάμε για τέτοιες προτάσεις θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι αυτό το οποίο θα κάνουμε δεν θα επηρεάσει αρνητικά την κοινωνική διάσταση από την ε, πλευρά των υπηρεσιών. Είναι προφανές ότι σε ορισμένες περιοχές της Ευρώπης θα υπάρξει βελτίωση διότι βλέπουμε ότι τώρα υπάρχει μία έλλειψη υποδομών και ιδίω όσον αφορά τις ενεργειακές επιλογές. Οι λύσεις θα πρέπει να είναι ε, ε, στη προσβάσιμες για τους καταναλωτές για να μπορέσουμε να έχουμε ε, μία ενιαία αντιμετώπιση. Ευχαριστώ. Τώρα από το Σουηδικό Ρίξτακ ο κύριος Περ Λέτλουντ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ για τόσες καλές και σοφές θα έλεγα παρεμβάσεις και προτάσεις στη συζήτηση. Είναι σαφές και για μας ότι θα πρέπει να μεριμνήσουμε, να διασφαλίσουμε αυτά τα πράγματα να γίνουν το δυνατόν ταχύτερα και να ληφθούν οι αναγκαίες αποφάσεις διότι η εμβέλεια αυτών των θεμάτων θα πρέπει να μας κάνει μέχρι το 2005 να εργαστούμε για να επιτευχθούν αυτά τα αποτελέσματα και φυσικά να χρησιμοποιήσουμε και τον ήλιο και το νερό, του υδάτινους πόρους, όλα αυτά για την επίτευξη της ενεργειακής αποδοτικότητας και να υπάρξει και η ενεργειακή διασύνδεση. Στην Σουηδία έχουμε το ε, ευτυχές γεγονός ότι έχουμε πολύ μεγάλο ποσοστό ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό η χρήση και η διασύνδεση των ηλεκτρικών δικτύων να επιτευχθεί. Αυτό θα έχει και το προτέρημα, το πλεονέκτημα να υπάρξει καλύτερη αντιστάθμιση σε σχέση με αυτές τις καλές πηγές ενέργεια Για παράδειγμα, όταν για παράδειγμα μπορούμε να εξαγάγουμε τις, ε, την ηλεκτρική ενέργεια που παράγουμε σε περιπτώσεις ε, ε, θετικής αιωλικής ενέργειας. Σε περίπτωση που κάτι αντίστροφο συμβαίνει θα μπορεί να εισάγεται η, ανα... η, ηλεκτρική ενέργεια που χρειαζόμαστε. Και έτσι διαπιστώνουμε ότι όλο και περισσότεροι πυρηνικοί αντιδραστήρες ε, δημιουργούνται, χτίζονται στην Ευρώπη. Δεν υπάρχει όμως ως προς αυτό μια πραγματική δυνατότητα για τον ανταγωνισμό. Υπάρχουν τόσα ανεπίλητα προβλήματα ακόμα τα οποία συνδέονται με τέτοιες πρωτοβουλίες. Αν υπάρξει ένα μεγαλύτερο ατύχημα στην Ευρώπη από πυρηνικούς αντιδραστήρες αυτό θα έχει πανευρωπαϊκές επιπτώσεις. Δηλαδή υπάρχουν προβλήματα για τα οποία δεν μπορεί μόνο μία χώρα να βρει τις λύσεις για αυτά Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό εμείς περιφερειακά τοπικά εθνικά να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και χρειαζόμαστε περισσότερα κονδύλια για μια τέτοια κατεύθυνση και ανάπτυξη αυτών των ε, ενεργειακών πηγών. Ένα πράγμα είναι απόλυτα σαφές, το ότι εμείς στην Ευρώπη θα πρέπει να κάνουμε μεγαλύτερη έρευνα για να μπορέσουμε να προωθήσουμε αυτές τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να επιτευχθεί το super grid, η μεγάλη διασύνδεση. Ε, Σας ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα η κυρία Μεντρισέβα που εκπροσωπεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κύριε Μάρια Ρίμπα, αγαπητοί συνάδελφοι, σήμερα χρειαζόμαστε μία πραγματική πολιτική ενεργείας και οι τελευταίες κρίσεις μας το υπενθυμίζουν η εγγύηση ε, μπορεί να μεταφραστεί σε ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η επάρκεια αυτή θα επιτευχθεί αν έχουμε καλύψει τα νότα μας στο εσωτερικό και στο εξωτερικό της Ενώσεως. Όσον αφορά το εσωτερικό θα πρέπει τα κράτη να συντονίσουν τις πολιτικές τους και ε, να επιτύχουν ένα καλύτερο σύντονισμό με περιφερειακές συνιστώσεις που θα μας επιτρέψει να διαφοροποιήσουμε και τις πηγές μας και τον τρόπο τροφοδοτήσεως. Θα επιτρέψει επίσης να βελτιωθούμε και γι' αυτό ο ρόλος των Εθνικών Κοινοβουλίων και η ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ τους θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη καλύτερη συνέπεια της νομοθετικής διαδικασίας και συντονισμό των κρατών μελών. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τις πολυμερείς σχέσεις και τις διμερείς σχέσεις αλλά θα χρειαστούμε μια πραγματική εξωτερική πολιτική ενέργεια και η Κάθριν Άστον θα πρέπει να αναλάβει την ευκαιρία που της δίδεται ώστε η υπηρεσία εξωτερικών σχέσεων να αποτελέσει το επίκεντρο το οποίο θα προβάλλει την κοινή πολιτική που θα έχουμε καταρτήσει όπως και τα μέτρα κατά τρόπο να υπάρχει συνεργασία μεταξύ κρατών μελών και μη κρατών μελών και φυστώ την προσοχή στη στρατηγική του Δούναβη που συνδυάζει συνεργασία κρατών μελών με μη Προφανώς δεν μπορούμε να είμαστε ουτοπιστές διότι τα κράτη-μέλη δεν θα απανηθούν τις ε, εξέχουσες σχέσεις που έχουν ίσως με ορισμένα κράτη εκτός ενώσεως αλλά θα πρέπει όλοι να ενταχθούμε στην κοινή πολιτική την οποία επιζητούμε και να καταρτήσουμε στα κείμενα ε, διατάξεις που θα επιτρέψουν καλύτερη τροφοδότηση και καλύτερα ε, δίκτυα. Θέλω να χαιρετήσω την παρουσία όλων των εθνικών βουλευτών σε αυτό το διήμερο διότι είναι ένα βήμα προς το εμπρός για μια κοινή πολιτική και σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι η συζήτησή μας ε, ε, μπορεί ε, να μεταδοθεί και εις τους πολίτες και έχουμε στον εξώστη ομάδες νέων και άλλο κρατήριο οι ευρωβουλευτές ε, ε, προσκαλούν ομάδες φιλοξενουμένων και ε, καλωσορίζω τους συμμετέχοντες που παρακολουθούν τη συζήτησή μας. Τώρα ο κύριος Τουσκέβιτς, ο οποίος εκπροσωπεί το Πολωνικό Κοινοβούλιο. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που μου δώσατε το λόγο και θα ήθελα να αναφερθώ σε συγκεκριμένα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε στην χώρα μου γύρω από θέματα όπως ε, η κατανάλωση της ενέργειας και η διαχείριση των αποβλήτων. Η διαχείριση των αποβλήτων είναι από τη φύση της μια διαδικασία ενεργοβόρα η οποία όμως θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή ενέργειας η βιομάζα σαν παράδειγμα για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος είναι μια γνωστή διαδικασία και νομίζω ότι θα πρέπει να στρέψουμε τις πιστώσεις που έχουμε στη διάθεσή μας στην ανακύκλωση, τη σωστή επιλογή των αποβλήτων, τον διαχωρισμό των αποβλήτων και την χρήση τους για παραγωγή ενέργειας. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να ιεραρχήσουμε σωστά τις επενδύσεις τις οποίες έχουμε διαθέσιμες στον συγκεκριμένο τομέα. Αυτό ήταν το πρώτο ε, κάπως συγκεκριμένο θέμα που ήθελα να σας θέσω. Το δεύτερο αφορά πάλι την διαχείριση των αποβλήτων αλλά σε τοπικό επίπεδο. Σαν παράδειγμα η λάσπη η οποία μπορεί να προέλθει από την ε, ε, διαχείριση των υγρών αποβλήτων είναι διαδικασίες όλες αυτές οι οποίες θα πρέπει να γίνονται σε τοπικό επίπεδο. Δεν θα πρέπει να υπάρχουν μεγάλες διαδρομές ε, ε, των αποβλήτων πριν την ε, αντιμετώπιση τους. Ο κ. Σκάβνο από το Ιρλανδικό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να μιλήσω λίγο για το θέμα της ασφάλειας στην προμήθεια ενέργειας και θα ήθελα να υπογραμμίσω αυτό το οποίο είπε και το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η σημασία της δικτύωσης δεν θα πρέπει να υποτιμηθεί. Και πέρυσι και φέτος τέσσερα δις δίδονται σε αυτούς τους τομείς για την βελτίωση των δικτύων και αυτό δεν είναι επαρκές. Μικρές χώρες σαν την Ιρλανδία, σαν τη δική μου, ε, προσπαθούν να γίνουν προς την Ευρωπαϊκή Ένωση εξαγωγής ενέργειας που προέρχεται από εναλλακτικές πηγές. Για να το πετύχουμε αυτό, απαιτείται θα έλεγα να υπάρξει καλύτερη διαδικτύωση. Θα πρέπει λοιπόν όλα αυτά τα θέματα να τα αντιμετωπίσουμε από κοινού, να καθορίσουμε έναν, όπως θα έλεγα, οδικό χάρτη, που θα επιτρέψει στις χώρες να προωθήσουν την παραγωγή τους εκεί όπου έχουν κάποια συγκριτικά πλεονεκτήματα. Σαν παράδειγμα αν είναι αποδεκτή ή μη πολιτική ή, ή μάλλον αν είναι αποδεκτή ή μη ατομική ενέργεια, αν έχουν οι χώρες μας κάποιες κλιματικές κάποια κλιματικά χαρακτηριστικά τα οποία μπορούν να βοηθήσουν. Μέχρι τώρα δεν έχουμε καταφέρει να ορίσουμε σωστά τα υπέρ και τα κατά των διαφόρων μορφών παραγωγής ενέργεια. Ενέργειας. Δεν έχουμε επίσης χρηματοδοτήσει σωστά τα δίκτυα τα οποία θα βοηθήσουν να συνδεθούν όλες οι περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ και 4-5 χρόνια ήμουν μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και είχα ζητήσει να υπάρξει ένα υπερδίκτυο είχα προτείνει να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιωλική στη θάλασσα. Ένα τέτοιο δίκτυο θα μπορούσε να τροφοδοτήσει σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό τις ανάγκες ε, όλων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα των παραθαλάσσιων. Λοιπόν, υπάρχουν επίσης θέματα ακόμα σε εκκρεμότητα σε σχέση με μονοπόλια, τα οποία εξακολουθούν να είναι ιδιοκτήτες και των δικτύων και ουσιαστικά να ελέγχουν και το σύνολο περίπου της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γύρω από το πρόβλημα αυτό. Και μια τελευταία παρατήρηση γύρω από τα βιοκαύσιμα κάθε χώρα αναπτύσσει τις δικές της πολιτικές και τις δικές της νομικές ρυθμίσεις γύρω από τα βιοκαύσιμα και την συμμετοχή τους ε, στην ε, βενζίνη και στο πετρέλαιο που καταναλώνεται από οχήματα. Αλλά δεν είναι σωστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση να χρησιμοποιούνται εντελώς διαφορετικά τέλη στήριξης των βιοκαυσίμων. Αυτές οι διαφορές αναχώρα νομίζω είναι αντίθετες με το πνεύμα και το γράμμα των κοινοτικών ρυθμίσεων. Ευχαριστώ πολύ κύριε Καβανό. Η κυρία Ζαλεύσκα από την Πολωνική ΣΕΙΜ. Θα ακολουθήσω ακριβώς συνεχίζοντας αυτά τα οποία ο συνάδελφος από την Ιρλανδία ανέφερε, διότι σε πολλές περιπτώσεις συμφωνούμε ή αναφέρουμε και τα εμπόδια, τα προσκόμματα στην υλοποίηση της κοινή ενεργειακής πολιτικής. Είναι λοιπόν θετικό παρόλα αυτά θα έλεγα αυτή η πρόταση διότι ταυτοποιώντας ε, τα εμπόδια και τα προσκόμματα μπορούμε να ακολουθήσουμε και να εκπονήσουμε μια κοινή στρατηγική. Η αηφορία και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν είναι μόνο η προστασία του περιβάλλοντος αλλά είναι και πολιτικός στόχος και αυτό τονίστηκε πολλές φορές στις συζητήσεις μας. Σημαντικό αυτό για να γίνει πιο ανεξάρτητη η Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τους ενεργειακούς πόρους. Αν όλα αυτά αληθεύουν. αν λοιπόν εξετάζοντας την κατάσταση σε διαφορετικές χώρες αυτό δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε σχέση με δυνατότητες ε, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν όμως δεν συγκλίνουμε τότε δεν θα υλοποιήσουμε τους στόχους υπέρ της προστασίας του περιβάλλοντος και δεν θα γίνουμε πιο ανεξάρτητοι. Στην έκθεση υπαριθμό 3 κάτι το οποίο τονίστηκε στη συζήτηση δεν αναφέρθηκε. Εγώ είχα τονίσει ότι δεν μπορούμε να μεταφέρουμε αυτόματα ενεργειακές λύσεις σε περιφέρειες σε ε, τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο με αυτόματο τρόπο. Αυτό αναφέρθηκε και από τον συνάδελφο από την Ιρλανδία, όπου οι γεωγραφικές συνιστώσεις καθιστούν ε, ανέφικτο ή δύσκολο το να επιτευχθεί αυτός ο ενεργειακός πόρος. Αυτό είναι σημαντικό. Επίσης υπογραμμίσαμε ότι η ευθύνη μας και η εγγύηση να έχει επιτυχή έκβαση η επένδυσή μας στους ενεργειακούς πόρους πρέπει να αναφέρεται πάντα στην προστασία των καταναλωτών και των συμφερόντων τους. Ιδιαίτερα σημαντικό για περιόδους κρίσης. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ για αυτά που είπατε. Εκπρόσωπος στη συνέχεια της Ιταλικής Γερουσίας θα λάβει τον λόγο. Άκουσα τις τρεις παρουσιάσεις από τις ομάδες εργασίας και θα ήθελα να σταθώ λίγο στην τρίτη ομάδα εργασίας να μου επιτρέψετε να κάνω εδώ κάποιες παρατηρήσεις. Σημερίζομαι τις παρατηρήσεις που έγιναν για τους δύο πρώτους πυλώνες της ανταγωνιστικότητας και της ασφάλειας έχω όμως κάποιες αμφιβολίες και τις εξέφρασα χθε στην ομάδα εργασίας για την ε, αντιμετώπιση ε, του, της παραγωγής ε, της εκπομπής καυσαερίων σαν δίκτυ παραγωγικότητας. Τώρα η Ευρώπη όπως είπα επηρεάζει κατελάχιστο κατελάχιστον παγκόσμια της ανθρωπογενείς εκπομπές καυσαερίων. Νομίζω ότι αυτό δεν φτάνει να το πούμε βέβαια. Θα πρέπει να προσθέσουμε στο κριτήριο της χαμηλής ή χαμηλότερης εκπομπής καυσερίων το θέμα, το πρόβλημα της εκπομπής χημικών ουσιών. Αυτό είναι το πρόβλημα το οποίο δημιουργεί τεράστιες συνέπειες στο περιβάλλον και στην υγεία των πολιτών. Έχουμε υπερεκτιμήσει το διοξίδιο του άνθρακα, τις παραδοσιακές δηλαδή εκπομπές καυσαερίων και υποτιμήσει τις χημικές ουσίες οι οποίες εκπέμπονται. Γενικά υπάρχει σοβαρό πρόβλημα σε σχέση με την παραγωγή αυτών των ουσιών. Ένα άλλο θέμα το οποίο θα ήθελα να υπογραμμίσω εδώ είναι η εξοικονόμηση ε, ενέργειας. Όταν χρησιμοποιούμε τον όρο αποτελεσματική χρήση της ενέργειας, τότε ναι, ε, εξοικονομούμε σβήνοντας τα φώτα, ε, εξοικονομούμε ε, ουσιαστικά μειώνοντας τις παραγωγικές μας δυνατότητες. Όχι, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τις παραγωγικές μας δυνατότητες με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και όχι απλά να βάζουμε μπροστά τη λέξη εξοικονόμηση. Ένα άλλο στοιχείο είναι ότι η προσπάθεια μείωσης του διοξιδίου του άνθρακα ε, θα πρέπει επίσης ε, να συνοδευτεί από αντίστοιχες προσπάθειες και άλλων χωρών στον κόσμο, γιατί αλλιώς θα έχουμε απώλειες οικονομικού τύπου. Θεωρώ επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να περάσει σε μια χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας με τον βέλτιστο κάθε φορά τρόπο. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα βελτιώσει συνηλικά την αποτελεσματικότητα του συστήματος. Ευχαριστώ πολύ για τη δήλωσή σας. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ως μέλος της Ευρωπαϊκή Συντακτικής συνέλευση. Ε, θυμάμαι πόσο μας ενδιέφερε να προσεγγίσει η Ευρώπη τους πολίτες. Και μας ενδιέφερε επίσης και η ενεργειακή ασφάλεια. Γι' αυτό θέλω να ευχαριστήσω για αυτή την ευκαιρία που μας δίνετε. Να κάνουμε λόγο για αυτά τα θέματα εδώ και να τα συζητήσουμε από κοινού. Σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα να συζητηθεί το θέμα της ε, οικοδόμησης της ευρωπαϊκής ε, κοινοτικής ενεργειακής πολιτικής ε, που είναι αναγκαίο στοιχείο για μας αν θέλουμε να καταδείξουμε την αλληλεγγύη και να εκφράσουμε αλληλεγγύη ο ένας προς τον άλλο. Κάνουμε λόγο για μια μακροπρόθεσμη προοπτική εδώ για αυτά τα οποία αφορούν νέες πηγές ενέργειας, διαφοροποίηση των πηγών, διασύνδεση και δυνατότητες διασύνδεσης ανεξαρτησία και ανεξάρτητες πηγές. Ε, φυσικά μην ξεχνάμε και την προστασία του περιβάλλοντος και την αποτελεσματικότητα όταν έρχεται η ώρα να κάνουμε λόγο για μηχανισμούς για την online απάντηση τις απαντήσεις online όσον αφορά τις απειλές που μπορούν να αναφύονται για τα ενεργειακά θέματα. Θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα στους φιλοξενουμένους μας, στον κύριο Πέδρο Λουίς Ματίνου Ρίβε και τον αντιπρόεδρο επίσης της Ευρωπαϊκής επιτροπή τον κύριο Χωακίν Αλμούνια. Κάναμε λόγο για τη συνθήκη της Λισαβόνας. Ξεκίνησαμε αυτό στην αρχή. Το ερώτημα είναι, οι διατάξεις ε, στην ε, συνθήκη της Λισαβόνας επακούν. Εχθέ, κατά τη διάρκεια τη προκαταρκτική τη πρώτη μα συνεδρίαση, ο πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κ. Γέζιο Μπούζεκ, ανέφερε ότι ίσω υπάρχει ανάγκη να καθελκίσουμε, να ξεκινήσουμε μια νέα χάρτα δικαιωμάτων και ένα ελάχιστο σύνολο υποχρεώσεων και καθηκόντων οι επαΐοντες, οι πραγματογνώμονες μιλούσαν, έκαναν λόγο για μια νέα δυνατότητα από πλευρά συνιστώσας τη συνθήκη για να εμβαθύνουμε στη συνέχεια τη συνεργασία μα στο ενεργειακό πεδίο. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν κάποιοι φόβοι. Αναφέρθηκαν από τον Πιέρ Λαγκιγέ. Το ερώτημα λοιπόν το οποίο αναφύεται είναι αν τα προβλήματα τα οποία συνδέονται με την υλοποίηση της συνθήκης της Λισαβόνας, αν τα προβλήματα αυτά δεν θα επαναληφθούν αν είναι, αν έρθει η ώρα και ακολουθήσουμε μια προσέγγιση υιοθέτηση μιας νέας συνθήκης ή νέας συνιστώσας συνθήκης, ερώτηση, χρειαζόμαστε κάποιες νέες λύσεις. Η πείρα μας δείχνει ότι δεν είναι μόνο οι διατάξεις και πάσης φύσεως έγγραφα τα οποία είναι σημαντικά, αλλά εκείνο το οποίο είναι το πιο σημαντικό είναι η πράξη, η δράση που επακολουθεί. Εμείς βιώσαμε μια κατάσταση όπου είχαμε εξαιρετικέ διατάξεις αλλά δεν υπήρχε δυνατότητα δράσης και τίποτα δεν λειτουργήσε καλά. Πρόεδρο σας ευχαριστώ καλά πολύ για αυτή την ε, δήλωση. Κύριος Σέρφ Προνιάρα από την Γαλλία παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πήραμε πολλές πληροφορίες από όλους τους εμπειρογνώμονες που είχαν προσκληθεί, που είχατε προσκαλέσει μας έδωσαν τις δυνατότητες να σκεφτούμε τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να ενισχύσουμε την συνεργασία της, ε, των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι παρεμβάσεις που έγιναν και στις ομάδες εργασίας και αυτές που ακούσαμε σήμερα το πρωί είχαν ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Βέβαια οι καταστάσεις που επικρατούν στο εσωτερικό των διαφόρων κρατών μελών ε, είναι εντελώς διαφορετικές. Προφανώς θα πρέπει να δώσουμε κάποιες προτεραιότητες στις ενέργειες που δεν παράγουν ε, ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα καυσαερίων και θα πρέπει να δούμε ακριβώς τι γίνεται και με τις μεθόδους ε, αποθήκευσης των αερίων αυτών. Υπάρχει επίσης το θέμα της σύνδεσης των δικτύων από τη μία με την ασφάλεια προμήθειας από την άλλη. Υπάρχει το θέμα της ανταγωνιστικότητας όπως επίσης και της σωστής κατανόησης της λειτουργίας της αγοράς. Αυτό είναι σημαντικό και για τις επιχειρήσεις αλλά και για τους χρήστες. Νομίζω ότι υπάρχει μια κοινή επιθυμία, μια κοινή πολιτική βούληση για να συνδυάσουμε τις προσπάθειές μας στην αναζήτηση και στην έρευνα νέων τεχνολογιών τεχνολογιών οι οποίες να καλύπτουν το σύνολο των διαθεσίμων μορφών ενέργειας όπως επίσης και το θέμα της αποθήκευσης της ενέργειας. Δεν αναφερθήκαμε ιδιαίτερα σε αυτό. Όταν έχουμε αποτελεσματικά συστήματα αποθήκευσης ενέργειας νομίζω ότι αυτό θα είναι ένα ουσιαστικό συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με άλλες περιοχές του κόσμου. Δεν μιλήσαμε επίσης και για το αποδεκτό ή μη περιβαλλοντικά των δυνατοτήτων παραγωγής ενέργειας από την κοινή γνώμη. Όλα αυτά δεν μπορούμε να τα αγνοήσουμε και δεν πρέπει να κάνουμε διακρίσεις ανάμεσά τους. Όλα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Τελειώνοντας, θεωρώ ότι ο έλεγχος της ενέργειας σε όλα τα στάδια της θα μας οδηγήσει και σε μικρότερη κατανάλωση και σε κατανάλωση μορφών ενέργειας που δεν θα παράγουν φαινόμενα θερμοκηπίου και στην δυνατότητα να αντιμετωπίζουμε συγκυριακές κρίσεις. Σε επίπεδο ανταγωνιστικότητας η Γαλλία βρίσκεται στη φάση μεταφοράς στην εσωτερική ενωμητάξη της ε, του τρίτου πακέτου μέτρων και να επανέλθω σε αυτά τα οποία είπε ο Υπουργό κ. Σουρίμπε προηγουμένω, ότι το θέμα εδώ δεν είναι τόσο θέμα νομικών μέσων τα οποία έχουμε ή δεν έχουμε στη διάθεσή μα, αλλά θέμα χρηματοδότηση. Ιδιωτική χρηματοδότηση, δημόσιων επενδύσεων. Αυτό είναι το βασικό ερώτημα πέραν από τις νομικές ρυθμίσεις. Σας ευχαριστώ πάντω για την οργάνωση αυτής της συνάντηση την οποία προσωπικά βρήκα ιδιαίτερω ενδιαφέρουσα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πουανιό. Ευχαριστώ. Και τώρα εν ονόματι του Κοινοβουλίου της Λιθουανίας ο κύριος Στακεβίτσος έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η συζήτησή μας εχθές και σήμερα τόνισε την έλλειψη πολιτικής βούλησης που χρειάζεται για να υπάρξει μια κοινή ευρωπαϊκή αγορά και μια κοινή ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική. Ο πρόεδρος Μπούζα οργάνωσε αυτή τη ε, στιγμή σε μια πολύ κατάλληλη εποχή για να κινητοποιήσει την πολιτική θέληση κατά τρόπον ώστε η Ευρώπη να μπορέσει να καταστεί μία πραγματική κοινότητα στο θέμα αυτό. Και έθεσε και τους στόχους αυτής της ενεργειακής ε, ε, κοινότητος, μια κοινή ενεργειακή αγορά, πολιτική και ασφάλεια ενεργειακή. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια εκπροσωπούνται σε αυτή τη συνάντηση και θα πρέπει ε, να ε, μπορέσουν να κινητοποιήσουν αυτή την θέληση. Το δικό μας κοινοβούλιο της Λιθουανίας στηρίζει αυτή την κατάρτιση της κοινότητας και θα θέλαμε η συνάντησή μας να στείλει ένα ηχηρό πολιτικό μήνυμα όσον αφορά αυτή την πρωτοβουλία. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Ο επόμενος ομιλητής εκπροσωπεί την γερουσία της Τσεχίας, ο κύριος Μπις. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Θεωρώ ότι πρέπει να πω ότι κάθε χώρα προσπαθεί να επιλύσει το ενεργειακό της μείγμα κατά τέτοιον τρόπο ώστε να επιτύχει ένα συνολικό στόχο, δηλαδή να μειώσει ε, το φαινόμενο του θερμοκηπίου και ε, να έχει και ένα καλό αποτέλεσμα. Εμείς δυστυχώς στη χώρα μας δεν έχουμε ούτε θάλασσα, ούτε ε, πολύ ε, αέρα, ούτε επαρκή ηλιοφάνεια, ούτε μπορούμε να έχουμε επαρκής ε, επερκέπω από θέματα βιομάζας γι' αυτό και ε, θεωρήσαμε ότι η πυρηνική τεχνολογία ε, δεν εκπέμπει οξύδιο του άνθρακος και μπορεί να έχει χαμηλές εκπομπές και μου έκανε εντύπωση αυτά τα οποία είπε ο εκπρόσωπος της Σουηδίας που έχει μεγάλη πείρα με τους πυρηνικούς αντιδραστήρες δεν πρέπει να φοβίζουμε τον κόσμο καταφερόμενοι κατά της ε, πυρηνικής ενεργείας. Αυτό δεν είναι σωστό και όσοι δεν πιστεύουν στην πυρηνική ενέργεια και ε, προκαλούν ε, αμφισβητήσεις για την ύπαρξη του φαινομένου του θερμοκηπίου ε, δεν θα συμβάλλουν εις την μείωση των εκπομπών και πιστεύω ότι ουσιαστικά κατά αυτόν τον τρόπο και με αυτές τις δηλώσεις δεν κάνουμε τις σωστές δηλώσεις και δεν θα επιτύχουμε το στόχο μας. Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, αν τώρα έχετε ερωτήσεις, παρακαλώ να σηκώσετε την μπλε κάρτα που σας έχει δοθεί. Ο συνάδελφος από την Ελλάδα και ο κύριος ε, ο, ο κύριος ήδη ε, έχει κάνει την ερώτησή του. Όποιος άλλος έχει μια ερώτηση προς όλους τους ομιλητές παρακαλείται να σηκώσει την κάρτα του και θα προσπαθήσω να σας δώσω το λόγο. Ε, συνάδελφε, για 30 δευτερόλεπτα. Θα ήθελα να σχολιάσω και να θέσω ένα ερώτημα για αυτά τα οποία άκουσα από τον τελευταίο μιλητή. Η Ευρώπη είναι όλο και περισσότερο μια ενιαία αγορά. Θα πρέπει να καταλήξουμε σε μια ευρωπαϊκή κοινότητα ενέργειας. Απαιτούνται δηλαδή και εδώ οδηγίες και κανονισμοί. Γιατί να μην αρχίσουμε λοιπόν να χρησιμοποιούμε την έννοια της εκπομπής καυσαερίων κατά κεφαλήν. Είναι κάτι το οποίο θα μας επιτρέψει να μετρήσουμε με πιο σωστό τρόπο τον περιορισμό της εκπομπής καυσαερίων και να καταστήσουμε και πιο ευαίσθητους στο πρόβλημα τους πολίτες της Ένωσης. Παρακαλώ πριν λέτε αυτά τα οποία είπατε να λέτε και το όνομά σας Λέγομαι Ρομπέρτο Τόρτολι από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Ιταλικής Δημοκρατίας. Παρακαλώ εσείς έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Σεσίλια Τσέντσετο από το Σουηδικό Κοινοβούλιο Ρίξτατ Έχω μία ερώτηση σε σχέση με την σουηδική τοποθέτηση όσον αφορά τα θέματα πυρηνικής ενέργειας. Στις 17 Ιουνίου θα γίνει ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο μας όπου θα πρέπει να λάβουμε απόφαση αν θα συνεχίσουμε με την εκμετάλλευση της πυρηνικής ενέργειας και θα δημιουργήσουμε νέους πυρηνικούς αντιδραστήρες ή όχι. Ο συνάδελφος ο προλαλής σας και εγώ συνεργαζόμαστε, εργαζόμαστε σε αυτό το επίπεδο. Δεν έχουμε υποχρεωτικά κάποια συνενετική ομόφωνη άποψη για το μέλλον και για τη Σουηδία είναι μια εναλλακτική λύση η πυρηνική ενέργεια ακόμα. Ευχαριστώ. The next speaker, please present Σας ευχαριστώ κυρία. Ο επόμενος ομιλητής να παρουσιαστεί και να αυτός συστηθεί. Φιλίπ Φορτελιέ, ε, Γάλλος ε, βουλευτής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όταν βλέπουμε το ποσοστό της τεχνικής φορολογίας ή στην τιμή της ενεργείας, μήπως ήδη δεν πρέπει να εκπονήσουμε μία φορολογική εναρμόνιση γιατί θα προσκρούσουμε σε αυτό το πρόβλημα για να δημιουργήσουμε μία ε, ενιαία αγορά ενεργειακή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Το επόμενο ερώτημα, εσείς κυρία μου. Χριστιανά Μπρούνερ από το Αυστριακό Κοινοβούλιο. Έχω να κάνω μία ερώτηση ε, σε αυτούς οι οποίοι θεωρούν την πυρηνική ε, ενέργεια σαν ε, κλιματολογική λύση. Για πόσο χρόνο πιστεύετε ότι θα είναι ακόμη η πυρηνική ενέργεια μία λύση και πιστεύετε ότι αξίζει να επενδύσει κανείς μεγάλα ποσά για αυτήν την ενέργεια αντί να τα χρησιμοποιήσει Εκτό εκτός από τις βασικές επιφυλάξεις που μπορεί να έχει, μπορεί να έχει κανείς για την ε, πυρηνική ενέργεια. Ευχαριστώ. Έχετε άλλες ερωτήσεις. Ίσως θα είναι ε, ερωτήσεις προς συναδέλφους που, είναι, που κάθονται στην αίθουσα. Μπορεί να έχουμε και μία συζήτηση από αυτού το επίπεδο. Ευχαριστώ. Εσείς ε, είμαι από το Βουλγαρικό Κοινοβούλιο και θέλω να κάνω μία ερώτηση. Πιστεύετε ότι μετά ε, από τη δημιουργία ενός ε, ενιαίου ευρωπαϊκού δικτύου, τη δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς και την εισαγωγή ανανεωσίμων πηγών ενεργείας θα μπορέσουμε να ε, συμπληρώσουμε και με άλλες ενέργειες όπως παραδείγματος ε, χάρη ε, όπου δεν υπάρχει ολική ενέργεια. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, Βίτμαν από το Αυστριακό Κοινοβούλιο. Για τους ε, Αυστριακούς το θέμα είναι που η Ευρώπη επενδύει στην πυρηνική ενέργεια, δηλαδή συνθήκη Ευρατών. Ε, αυτό το ποσό προς το πνεύμα το οποίο συζητήσαμε, δηλαδή ένα δισεκατομμύριο ευρώ για την Αυστρία θα μπορούσε αντί να χρησιμοποιηθεί για την ατομική ενέργεια να χρησιμοποιηθεί χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη ανανεωσίμων ενεργειών. Ευχαριστώ. Υπήρξαν και κάποιες ερωτήσεις που είχαν σχέση με, τα πυρηνικά, με τους πυρηνικούς σταθμούς όπου υπάρχουν αντιφατικές απόψεις. Μήπως κάποιος ε, θέλει να απαντήσει ε, σχετικά με την πυρηνική ενέργεια. Ε, δηλαδή τι θα έπρεπε να γίνει. Ε, η απάντησή σας μπορεί να καλύψει ένα λεπτό. Ε, θέλω να κάνω μία ερώτηση προς τον Σουηδό συνάδελφο. Τι θα γίνει στην περίπτωση όπου η υπερθέρμανση του πλανήτη φτάσει σε υψηλά επίπεδα με όλα αυτά τα πυρηνικά εργοστάσια τα οποία προτείνεται. Well, uh, uh, Συνάδελφοι, θα ήθελα να ρωτήσω. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση σχετικά με την πυρηνική ενέργεια και είναι ευθύνη του κάθε κράτους μέλους να αποφασίσει τι ενεργειακό μείγμα θέλει να επιτύχει. Ε, ξέρουμε ποια είναι τα κίνητρα, ξέρουμε ποιες είναι οι ανάγκες ε, για την ε, περιβαλλοντολογική προστασία και δεν αναφέρομαι μόνο στο κλίμα αλλά και το περιβάλλον με τα απόβλητα, την σκόνη οπότε δεν πρέπει να επικεντρωθούμε σήμερα σε αυτό το συγκεκριμένο πρόβλημα. Ας το αφήσουμε ως έχει στη διάκριση των κρατών μελών και ίσως ε, για σήμερα αυτή είναι η καλύτερη λύση. Και τώρα θα ήθελα να δώσω τον λόγο. Ελπίζω ότι η ερώτησή σας δεν έχει σχέση με την πυρηνική ενέργεια. Εντάξει. Ήθελα απλώς να σας πω ότι συμφωνώ με την άποψή σας. Ευχαριστώ. Καταρχήν και εγώ θα ήθελα να συμφωνήσω με την παρατήρησή σας, αλλά έχω μία ερώτηση και θα ήθελα να θίξω και ένα άλλο θέμα ε, διότι αν γίνει αυτή η συζήτηση θα πρέπει η συζήτηση να γίνει με το να, να τεθεί το ερώτημα τι ε, λύσεις υπάρχουν και νομίζω ότι οι λύσεις είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Πιστεύω ότι αυτό είναι αδιαμφισβήτητο. Εκτός όμως από την βιομάζα που έχει διάφορα άλλα προβλήματα ε, <clears throat> υπάρχουν επιπλέον δύο ουσιαστικά άλλα προβλήματα Καταρχήν, ε, ότι είναι θέμα μεγέθους και θα πρέπει να υπάρξει αποθήκευση διότι οι ανανεώσιμες πηγές ενεργείας για να μπορέσουν να συμμετέχουν περισσότερο θα πρέπει να μπορούν να αποθηκευτούν και αναφέρομαι εδώ στα υδροελεκτρικά προγράμματα που πρέπει να βελτιωθούν και επίσης Ελπίζω ότι ε, θα μπορέσουμε να αποφύγουμε ε, τα ατυχήματα. Ε, δεν είχαμε σημαντικά ατυχήματα σε υδροελεκτρικά έργα τα τελευταία χρόνια, αλλά μην ξεχνάμε τι μπορεί να συνεπιφέρει ένας σεισμός. Επίσης, όσον αφορά την, τον ηλεκτρισμό, όπως είπα και χθε, το μικρότερο τμήμα είναι ο ηλεκτρισμός όσον αφορά πηγές ενέργειας. Το χειρότερο είναι ε, η κινητήριος δύναμη. Ευχαριστώ και ε, τώρα ε, τελευταία συζήτηση ξεκινά και απαντήσεις θα ξεκινήσει ο κύριος Μαρίν Ουρίβε που έχει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ για όλες αυτές τις παρεμβάσεις που ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσες και επικοδομητικές για την ευρωπαϊκή αυτή συζήτηση των θεμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο των ενεργειακών θεμάτων. Κάποια σύντομα σχόλια θα ήθελα να κάνω ολοκληρώνοντας. Πρώτα απ' όλα, <clears throat> υπάρχει εγγενή ανησυχία όσον αφορά την ασφάλεια και την ασφάλεια του ανεφοδιασμού. Είναι ένα λογικό, μια λογική μέρημνα αυτή. Παραδοσιακά είχαμε υψηλότατη εξάρτηση που βρίσκεται στο 60% για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε πολλές χώρες αυξάνεται και φτάνει ως το 80% αυτή η εξάρτηση. Και εδώ έχουμε το θέμα των πρώτων υλών, όπως είναι το φυσικό αέριο. Και τα προβλήματα αυτής της εξάρτησης καταδείχθηκαν ανάγλυφα με πολύ χαρακτηριστικό τρόπο πέρυσι όσον αφορά τον ανεφοδιασμό με φυσικό αέριο. Πράγμα το οποίο έτυχε της προσοχής όλων των χωρών και έδειξε ποια είναι η κατάσταση με την εξάρτηση από έναν πάροχο ενεργειακού πόρου για το φυσικό αέριο το να εξαρτώμαστε σε τόσο υψηλό βαθμό από την, τον ανεφοδιασμό μας από ένα παρόχο μπορεί να είναι ένα ενδυνάμει όχι μόνο θεωρητικά πρόβλημα αλλά και πραγματικό μεγάλο πρόβλημα και γι' αυτό το πρόβλημα της ασφάλειας ανεφοδιασμού έχουμε τον στόχο της δημιουργίας μιας πραγματικής ενιαίας εσωτερικής αγοράς ενεργειακών πόρων που θα μας δώσει τη δυνατότητα να πολυμορφοποιήσουμε την εξάρτησή μας από αυτούς τους πόρους. Διότι αν αληθεύει ότι αυτή η εξάρτηση φτάνει το 80% σε κάποιες χώρες, η εξάρτηση από έναν και μόνο φτάνει για κάποιες χώρες 100%. Αυτά είναι τα στοιχεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο που είναι ανησυχητικά και έτσι λοιπόν πρέπει να δούμε μια πρώτη απάντηση από πλευρά μα που είναι αυτή. Άλλε απαντήσει είναι η υποκατάσταση με ε, αυτή το αυτογενείς ε, ε, επιτόπιους πόρους, ε, ενεργειακούς πόρους. Κατά τη διάρκεια της Ισπανικής Προεδρίας είχαμε ως μία από τις προτεραιότητές μας την ασφάλεια του ανεφοδιασμού στους ενεργειακούς πόρους. Προχωρήσαμε εγκρίνοντας ένα κανονισμό όσον αφορά τις επενδύσεις στο Συμβούλιο του Μαρτίου που δίνει προβλεψιμότητα μεσοπρόθεσμα. Προχωρήσαμε πολύ και θέλω να ευχαριστήσω δρατώμενος ευκαιρίας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τον επικοδομητικό διάλογο που διαμόρφωσε κατά τη διάρκεια αυτή τη περίοδου. Προχωρήσαμε έτσι όσον αφορά τον κανονισμό για τον ανεφοδιασμό με φυσικό αέριο και ελπίζουμε ότι μπορούμε να ολοκληρώσουμε τη διαπραγμάτευση κατά τη διάρκεια αυτού του εξαμήνου σε συνεργασία πάντα με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επίση, διοργανώσαμε μια διάσκεψη για τι υποδομέ για να διευκολύνουμε την επίτευξη αυτού του μέσου στι υποδομέ αυτού που θα προτείνει κατά τη διάρκεια του δεύτερου εξάμεινου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εξετάζοντας όλες τις μορφές και τρόπους δράσης και συνεργασίας με τρίτες χώρες όσον αφορά την ασφάλεια ανεφοδιασμού σε ενεργειακούς πόρους. Αλλά σίγουρα ένα θέμα που χωρίς αμφιβολία παραμένει πολύ σημαντικό είναι το θέμα της χρηματοδότησης. Το ανέφερε ο κύριος Πονιάν η χρηματοδότηση των υποδομών. Σίγουρα οι υποδομές είναι μία από τις πτυχές εκείνες όπου πολλές φορές εκείνοι οι οποίοι υφίστανται από τις επιπτώσεις για τις υποδομές δεν είναι αναγκαστικά εκείνοι που εποφελούνται περισσότερο. Υπάρχει και μια εξωτερική συνιστόσα για τους υπόλοιπους. Και αυτό δίνει τα μέσα της αγοράς τα οποία δεν λειτουργούν πάντα τέλεια. Γι' αυτό χρειάζεται μια παρέμβαση. Μια παρέμβαση στην υποστήριξη των προγραμμάτων και σχεδίων διευκολύνοντας κάποια βήματα. Υπάρχουν ευρωπαϊκοί στόχοι ακόμα και επίτευξη του 10% μεταξύ των κρατών μελών και είχαμε και συζήτηση με τον Επίτροπο για τα θέματα ενέργειας στη Μαδρίτη, είναι ακριβώς ένας από τους στόχους που δεν πετύχαμε αποτύχαμε τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πετύχουμε να υλοποιηθούν αυτοί οι στόχοι. Και έλεγα ότι ένας από τους μεγάλους στόχους που απέμενε είναι η αξιοπιστία της επίτευξης αυτών των στόχων. Ενώ σε άλλους τομείς όπως ε, για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας <clears throat> προχωρούμε με καλούς ρυθμούς. Πρέπει να διασφαλίσουμε αυτή την αξιοπιστία, να την εξασφαλίσουμε αλλά και με τα χρηματοδοτικά μέτρα που απαιτούνται και μέσα που απαιτούνται να καθορίσουμε προτεραιότητες στις δράσεις μας. Έχουμε και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα για την Οικονομική Συνεργασία. Αυτά τα στοιχεία είναι <clears throat> συγκυριακά όμως περισσότερο. Χρειάζονται τα μέτρα υποδομών ώστε να υπάρξει διασφάλιση της χρηματοδότησης. Έγινε πολλή λόγος για μια δεύτερη πτυχή για την ενιαία εσωτερική αγορά. Έγινε λόγος για την διαφοροποίηση, διαχωρισμό της ιδιοκτησίας μεταξύ των ε, παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας και των ιδιοκτητών των δικτύων διανομής των ηλεκτρικών δικτύων. Έχουμε ένα πρότυπο unbundling με τρεις εναλλακτικές δυνατότητες που πρόσφατα εντάχθηκε στο πακέτο απελευθέρωσης, ευρωπαϊκής απελευθέρωσης και ελπίζουμε ότι θα μπορέσει από τα κρατη και έτσι να μπορέσει να λειτουργήσει ε, πολύ σύντομα. Με ρωτούσατε επίσης, με ρώτησε ο εκπρόσωπος της Ελλάδας, ο κύριος ε, ε, από την Βουλή των Ελλήνων, για την επίπτωση όσον αφορά την απελευθέρωση των τιμών. Νομίζω η επίπτωση δεν είναι το ότι θα υπάρξει υποχρεωτικά μια μείωση των τιμών, αλλά η απελευθέρωση θα επιτρέψει οι τιμές να αντανακλούν το κόστος των προϊόντων ως προϊόντων που συζητούμε. Λαμβάνοντας υπόψη ε, την ύπαρξη κάποιων προστατευόμενων πελατών ή ε, κάποιων ε, που θα πρέπει να προστατεύονται και αυτό επίσης εντάσσεται στο πακέτο μέτρων. Αλλά θα πρέπει η απελευθέρωση να αντανακλά το κόστος της παραγωγής, να δημιουργηθεί ένας ευρωπαϊκός χώρος με κανόνες παρόμοιους στις χώρες μας για να μπορούν να ανταγωνιστούν οι χώρες μας αναμεταξύ τους σε ένα αυθεντικά θεμητό πεδίο, για να υπάρχει ένα πεδίο ενεργοποίησής μας. Σε αυτό είναι σημαντικό και διασύνδεση. Είναι πολύ δύσκολο ε, προσπαθώντας να απελευθερώσει κανείς μικρές και απομονωμένες αγορές, μικρές, ε, μικρά νησιά. Η ε, κατάσταση αυτή δεν διευκολύνει την απελευθέρωση, διότι πολλές φορές θα δούμε μονοπόλια να υφίστανται εκεί, με πολύ μικρή δυνατότητα ανταγωνισμού. Δεν έχουμε λοιπόν έτσι την εγγύηση το κόστος να αντανακλά, οι τιμές να αντανακλούν το κόστος. Θα πρέπει να συνοδεύεται λοιπόν η προσπάθεια από αυτή την ενιαία εσωτερική αγορά για την οικοδόμησή της. Και αυτό είναι δυνατό να γίνει με την κινητοποίηση όχι μόνο κεφαλαίων, αλλά και την κινητοποίηση αγαθών, ενεργοποίηση και κινητοποίηση αγαθών για τα ενεργειακά θέματα. Αυτή η απελευθέρωση πρέπει να είναι ένα κίνητρο για την αποτελεσματικότητα, γιατί πρέπει να προσπαθήσουμε να πετύχουμε αυτή την αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων. περνώντα το θέμα τη αποτελεσματικότητας πρέπει να υπενθυμίσουμε την παρέμβαση που έγινε για το πώς θα μπορέσει να δράσει η αποτελεσματικότητα. Η αποδοτικότητα, η αποτελεσματικότητα είναι ένα στοιχείο κλειδί για τις, ε, τους στόχους μας. Για τους στόχους μας όσον αφορά την εκπομπή ρήπων, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ε, η αποδοτικότητα στην ενέργεια είναι ένας κοινό παρονομαστής. Όχι μόνο πρέπει να δημιουργούμε όλο και περισσότερο στις ε, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά να προσαρμόσουμε περισσότερο την κατανάλωση στις ανάγκες μας. Γι' αυτό η αποδοτικότητα πρέπει να είναι το κυριότερο μέσο με το οποίο η αποτελεσματικότητα αυτή θα δώσει τη δυνατότητα να πετύχουμε τους στόχους μας στο μέλλον στου ενεργειακού πόρου. και χωρί αμφιβολία την αποδοτικότητα δεν μπορούμε να την πετύχουμε μόνο λέγοντα στου πολίτε μα να εξοικονομούν ενέργεια και να καταναλώνουν λιγότερο. Πρέπει να στοιχηματίσουμε και να επενδύσουμε υπέρ των νέων τεχνολογιών που θα βελτιώνει την χρήση των ενεργειακών πόρων και θα δίνει τη δυνατότητα πιο ορθολογική εκμετάλλευση των ενεργειακών πόρων αλλά πάντα με την τεχνολογική ανάπτυξη νέων δυνατοτήτων. Επίση, θα ήθελα από την άλλη πλευρά να επικεντρωθώ στο θέμα των τεχνολογιών. Η τεχνολογία είναι μια άλλη μεγάλη πτυχή που χρειάζεται χρηματοδότηση. Όλοι γνωρίζουμε και αναγνωρίζουμε ότι οι τεχνολογικές πραγματικότητες είναι εκεί όπου υπάρχει η μεγαλύτερη έλλειψη νέων τεχνολογιών στις αγορές, όπου έχουμε ελλείψεις και δεν λειτουργούν τα πράγματα καλά. Υπάρχουν λοιπόν ε, θετικές πτυχές ε, που απορρέουν συνολικά για την οικονομία και εδώ ε, σε σχέση με την συμμετρία ε, ε, των δράσεων. Πρέπει η χρηματοδότηση να είναι ένα στοιχείο θεμελιώδες και έτσι να δράσουμε. Αυτό αντανακλάται και συμπεριλαμβάνεται στα συμπεράσματα που πρόσφατα υιοθέτησε το Συμβούλιο όσον αφορά το πρόγραμμα δράσης για τα επόμενα χρόνια. Επίσης συμπεριλαμβάνονται εδώ συμπεριλαμβάνεται η διάσκεψη για το set plan και οι διάφορες πρωτοβουλίες. Η τεχνολογία, όπως είπα και στην αρχική μου παρέμβαση, είναι κέρια σημασία στοιχείο. Κέρια σημασία στοιχείο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Όχι μόνο για να πετύχουμε αυτές οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας να είναι ανταγωνιστικές και να προσφέρονται σε προσιτές τιμές στους καταναλωτές. Είναι θεμελιώδης για να πετύχουμε τη σωστή διαχείριση αυτών των τεχνολογιών που ακριβώς έχουν δημιουργούν ένα πρόβλημα όχι αποθήκευσης ε, αλλά για το ότι θα πρέπει να δούμε πώς θα πρέπει να λαμβάνονται οι αποφάσεις για το τι θα πρέπει να παράγεται και πόσο. Μια διαχειρισιμότητα, ένα θέμα διαχείρισης το οποίο θα ήταν μικρότερο πρόβλημα αν είχαμε υψηλό επίπεδο διασύνδεσης διότι οι ροές σε σχέση με μεγάλο επίπεδο, υψηλό επίπεδο διασύνδεσης διευκολύνουν την υπόθεση. Χωρίς αμφιβολία όταν έχουμε μικρές αγορές με υψηλό αριθμό ανανεώσιμων πηγών ενέργειας λαμβάνουμε υπόψη όπως και στην στην ισπανική αγορά ότι για παράδειγμα για την αιωλική παραγωγή ενέργειας ε, που σε κάποιες ζώνες ε, ε, επιτυγχάνει ποσοστό 50% επίτευξης έχουμε όμως και το θέμα της, του βορρά και του νότου της ανατολής και της δύσης της επικράτειάς μας και σε μια χώρα σαν την Ισπανία ας δούμε το σύνολο τώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπου είναι μεγαλύτερες οι διαφορές μεταξύ βορρά που έχει αιωλική ενέργεια, ήλιου, ηλιοφάνεια στο νότο, στις νότιες χώρες. Ε, ε, αυτό το πρόβλημα της ε, διαχειρισιμότητας, της σωστής διαχείρισης που θέτει προβλήματα ήδη στις μικρότερες χώρες είναι, μπορεί να αντιμετωπιστεί επίσης και σε μεγαλύτερη κλίμακα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η τεχνολογία πρέπει να ληφθεί υπόψη και να ενταχθεί. Η ένταξη νέων τεχνολογιών στο δίκτυο. Ο κύριος από τη Βουλγαρία ρωτούσε πώς θα επιληθεί αυτό το πρόβλημα παράδειγμα στις χώρες όπου υπήρξε ανάπτυξη πολύ σημαντική των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καταδείχθηκε ότι είναι δυνατόν να ενταχθούν με συστήματα εφιούς διαχείρισης και με την αποτελεσματική διασύνδεση σε σχέση με την παραγωγή να γνωρίζουμε ακριβώς ε, τι θα χρειαστεί από πλευράς παραγωγής και με συστήματα αποθήκευσης, εναποθήκευσης ή και άλλα συστήματα τα οποία θα αναπτυχθούν τα επόμενα χρόνια και επί των οποίων εδράζονται και εργάζονται οι νέες, ε, ε, επικεντρώνονται οι νέες τεχνολογίες. Τεχνολογίες που θα κάνουν το backup, που θα μπορέσουν να καλύψουν τις ανάγκες και τα κενά, να είναι διαθέσιμες όταν θα χρειάζονται σε περιόδους εχμής και να μπορούν έτσι να καλύπτουν τα κενά με την ένταξη σε ένα δίκτυο. Στόχος και πρόκληση πάρα πολύ μεγάλη για ένα σύστημα το οποίο δεν έχει επιτύχει τον ε, ευκταίο βαθμό διασύνδεσης θα πρέπει να δούμε αυτή την πτυχή. Δεν θέλω να επαναλάβω το παράδειγμα της Ισπανίας που έχουμε κάποιες 50, ε, σε κάποιες περιοχές 50% παραγωγή ε, ηλεκτρικής ενέργειας από την αιωλική ενέργεια ε, σε περιόδους εχμής όταν χρειάζεται. Γι' αυτό λοιπόν η τεχνολογία θα πρέπει να δώσει τις απαντήσεις που χρειαζόμαστε. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σχολιάστηκε αληθεύει ότι επικεντρώνεται στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ε, συνολικά ως δράση. Όμως ε, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να είναι ένα από τα στοιχεία κλειδιά για το άμεσο μέλλον αν θέλουμε να πετύχουμε τους στόχους μας ε, σε σχέση με τα ανανεώσιμα πρέπει να δούμε ε, την ε, ε, κλιμακούμενη δράση και θα πρέπει περισσότερο να λάβουμε υπόψη αυτή τη συνιστόσα. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει να προχωρήσει. Το θέμα της κινητο... κινητικότητας, η δημιουργία και ανάπτυξη ηλεκτρικών οχημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό θα δώσει τη δυνατότητα ένταξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε ένα τόσο σημαντικό πεδίο. Πάνω από 50% της ενεργειακής κατανάλωσης. Και προφανώς αν δεν είμαστε στεναροί στην ανάπτυξή τους, πέρα από την ανάπτυξη ανάπτυξη και νέων καυσίμων θα έχουμε πολλά προβλήματα για την επίτευξη των στόχων μας πέρα από το 2020 υπό τους όρους εκπομπών ρήπων. Και τέλος, να αναφέρω τον ρόλο της τεχνολογίας ε, και πάλι στην διαχείριση των ενεργειακών θεμάτων. Δεν μπορούμε να ζητήσουμε να ε, σβήνουν, ε, τους, να κλείνουν τους διακόπτες. Πρέπει να υιοθετήσουμε ευφυή συστήματα χρήσης ενέργειας ώστε να μπορούμε στις ώρες μη εχμής να μπορούμε να να ε, δρούμε πιο αποτελεσματικά όταν, και όταν θα υπάρχει τότε μικρότερο κόστος ε, να μπορούμε με πιο ορθολογικό, πιο αποτελεσματικό τρόπο να εκμεταλλευόμαστε τη διαθέσιμη ενέργεια. Και ένα άλλο θέμα για τη σύλληψη και αποθήκευση διοξιδίου του άνθρακα. Μια και ε, τα ορυκτά καύσιμα θα συνεχίσουν στο άμεσο μέλλον να διαδραματίζουν ένα ρόλο, πρέπει να δούμε και αυτή την συνιστόσα αν θέλουμε να ανταποκριθούμε με τις υποχρεώσεις εκπομπών ρήπων στο περιβάλλον. Και η σύλληψη και αποθήκευση διοξιδίου του άνθρακα θα πρέπει να διαδραματίζει ένα ρόλο. Και αυτό μπορεί μόνο να γίνει με την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών. Επίση, ρώτησε ο κύριο Ρώση ποια είναι τα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσει μια συγκεκριμένη βιομηχανία ή αυτοκινητοβιομηχανία για παράδειγμα. Με αυτά τα στοιχεία υπόψη θα πρέπει να μπορέσουμε να δράσουμε ώστε να μπορούν να είναι ανταγωνιστικέ αυτέ οι βιομηχανίε μα. Αυτά θα έπρεπε να αναφέρω. Ολοκληρώνω την παρέμβασή μου με το σημείο εκείνο για το αν επαρκεί η συνθήκη Λισαβόνα για να πετύχουμε του στόχου μα ή όχι. Ένα στοιχείο κλειδί για τη συζήτηση και σήμερα και χθε στι συζητήσει. Εάν χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω. Νομίζω ότι τα λόγια του κυρίου Βέιτμπροντ από την Πολωνία όταν διατύπωσε αυτό το ερώτημά του στο συμπέρασμά του δίνουν ένα σημαντικό τμήμα της απάντησης. Αυτό που χρειαζόμαστε χωρίς αμφιβολία είναι η βούληση να δράσουμε, πολιτική βούληση. Δεν είναι πρόβλημα νομοθετικών μέσων και εργαλείων. Τώρα, για μια χάρτα δικαιωμάτων που θα αντανακλά αυτή τη βούληση, καλοδεχούμενη είναι μια τέτοια πρωτοβουλία. Όμως θα πρέπει να δούμε το θέμα της ε, ρύθμισης. Ε, αν ε, πρέπει να υπάρχει η βούληση η πολιτική και να αντανακλάται η πολιτική βούληση με αυτόν τον τρόπο που χωρίς αμφιβολία είναι πολύ σημαντικό στοιχείο σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να προχωρήσουμε. Να δώσει τα κλειδιά για την αηφορία και την ε, αποτελεσματικότητα προς όφελος των πολιτών μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για τις παρατηρήσεις σας. εκπροσωπήσατε την ε, Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τώρα θα δώσω το λόγο στον Αντιπρόεδρο Αλμούνια. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ λοιπόν δεν θα προσθέσω πολλά σχόλια σε αυτά τα οποία μόλις έκανε ο Υφυπουργός κ. Πέντρο Μαρίν, διότι συμπίπτω ουσιαστικά με όλα τα οποία προανέφερε και είπε απαντώντας στις παρεμβάσεις και στις ερωτήσεις που διατυπώθηκαν προς αυτόν. Όμως, αυτό που θα κάνω είναι θα επικεντρωθώ ιδιαίτερα σε κάποια λίγα σημεία. Πρώτα απ' όλα υπήρξε μια ερώτηση <clears throat> από πλευράς ε, ενός Ευρωβουλευτή που αναφερόταν άμεσα στο τι κάνει λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρησιμοποιώντας τα μέσα της πολιτικής για τον ανταγωνισμό σε σχέση με τον ενεργειακό τομέα. Αυτή ήταν η ερώτηση χωρίς να επισέθω στην συγκεκριμένη περιγραφή όλων και κάθε μιας από όλες αυτές τις δράσεις που είναι πολλές, αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι είναι πολύ σημαντικό. Σημαντική πρωτοβουλία που υιοθέτησε η συνάδελφός μου Νέλη Κρούς κατά τη διάρκεια της προηγούμενης Επιτροπής να γίνει μια σφιγμομέτρηση sector, sector inquiry για τον τομέα του, της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου. Μια ανάλυση σε βάθος και κινώντα από τις ε, πληροφορίες που είχαμε επιτόπου στη διάθεσή μας. Δηλαδή επιτόπου με επισκέψεις στις, ε, ε, στο εσωτερικό των επιχειρήσεων και βιομηχανιών σε πολλές από αυτές. Αυτή η σφιγμομέτρηση sector inquiry Έδωσε τη δυνατότητα άμεσα από πρώτο χέρι να πάρουμε στοιχεία, γνωρίζοντας τα στοιχεία αιτίου και αιτιατού, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε προβλήματα δεσπόζοντος ρόλου, προ, πρακτικές στρέβλωσης του ανταγωνισμού σε πολλές ε, περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα <clears throat> δεν αφαιρόμαστε εδώ μόνο στις, ε, σε άγνωστες, κάποιες άγνωστες επιχειρήσεις, αλλά στην Electricité de France, για παράδειγμα, EDF, την E.ON στη Γερμανία, <clears throat> για να αναφέρω δύο μεγάλες ε, ε, εταιρείε παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Υπάρχουν τοποθετήσεις και δράσεις σαν συνέπεια αυτής της μελέτης αυτού του τομέα. Inquiry ε, sector Inquiry. Αλλά επίσης αυτή η μελέτη έδωσε την δυνατότητα στην Επιτροπή τότε να θεμελιώσει καλύτερα, να βασίσει καλύτερα και να επικεντρώσει με καλύτερο τρόπο τις προτάσεις της για το τρίτο νομοθετικό πακέτο, πακέτο μέτρων για τα ενεργειακά. Αυτή η δράση λοιπόν που είναι ένα πρότυπο το οποίο υλοποιήθηκε επίσης και σε άλλους σημαντικούς τομείς για τη λειτουργία Τη ενιαία εσωτερική αγορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως είναι τα φαρμακευτικά προϊόντα και σκευάσματα ή δραστηριότητε όσον αφορά το χρηματοπιστωτικό τομέα, τον τραπεζικό τομέα, στο λιανικό εμπόριο, retail. Είναι πολύ σημαντικέ δράσει όσον αφορά τα θέματα ανταγωνισμού που στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτού του ενεργειακού τομέα για την ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο αποτέλεσαν βάση και δίνουν βάση για συγκεκριμένες χειροπιαστές αποφάσεις από πλευράς μας. Και επιπλέον δρούμε με διαρκή χαρακτήρα επιτηρώντας την υλοποίηση των υποχρεώσεων όσον αφορά τις επιχορηγήσεις, κρατικές ενισχύσεις. Στο θέμα των κρατικών ενισχύσεων έχει ανοίξει η συζήτηση σήμερα και τώρα για το πώς θα ενταχθούν στην δική μας προσέγγιση της συμβατότητας ή όχι με τους γενικούς κανόνες όσον αφορά τις επιδοτήσεις και των μέτρων που θα λειτουργήσουν ή θα δρομολογηθούν για την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών. Υπάρχει εδώ μια σημαντική συζήτηση για τον τρόπο με τον οποίο υπό το πρίσμα του ελέγχου και της εποπτείας των κρατικών επιδοτήσεων και ενισχύσεων θα μπορέσουμε να εργαστούμε και να συνεργαστούμε να δούμε πώς θα διαμορφωθούν τα δικαιώματα εκπομπών ρήπων ώστε με το σύστημα αυτό εκκυρώνοντας από το 2013 αυτά τα ε, δικαιώματα ε, εκπομπών ρήπων να μην χορηγούνται δωρεάν στο πρωτογενή τομέα εκπομπών αλλά να γίνονται πληστηριασμοί να ε, εκποιούνται ώστε εκεί όπου υπάρχει μεγάλη ενεργοβόρα ας το πω έτσι δράση θα χρειαστεί ειδική αντιμετώπιση ώστε να αποφύγουμε αυτή η τομείς σαν συνέπεια των επιβαρύνσεων που θα σημαίνει ένα νέο σύστημα εμπορίας εκπομπών ρήπων για την παραγωγή και εκπομπή διοξιδίου του άνθρακα στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση να μην έχουν τον πειρασμό να μεταβούν, να μετεγκατασταθούν αλλού εκεί όπου δεν θα υπάρχουν δεσμεύσεις παρόμοιες με αυτού του νέου συστήματος και να συνεχίσουν να εκπέμπουν λοιπόν διοξίδιο άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Πρέπει να αποφύγουμε αυτή την μετεγκατάσταση από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε περιοχέ που δεν θα υφίστανται αυτού τους περιορισμούς είναι μια συζήτηση πάρα πολύ σημαντική που έχει ξεκινήσει και που πρέπει να αντιμετωπιστεί και να επιληθεί παράλληλα με τη συζήτηση και τη διαπραγμάτευση που είναι ακαθόδης για αυτό το νέο σύστημα μετά το Κιώτο, για την περίοδο μετά το Κιώτο. Είδαμε στη Σύνοδο της Κορυφής της Κοπενχάγης ότι δεν είναι εύκολο να προχωρήσουμε, να εντάξουμε εκείνους που δεν είχαν ενταχθεί στο πρωτόκολλο του Κιώτο σε ένα συνεκτικό πλαίσιο. Υπάρχει πολλή δουλειά λοιπόν για όλα αυτά που πρέπει να γίνει για τα ε, μέσα της πολιτικής για τον ανταγωνισμό και τη σωστή λειτουργία τους για την αντιμετώπιση του προβλήματος του δεσπόζοντος ρόλου και την αντιμετώπιση των προβλημάτων καρτέλ και μονοπωλίου και το θέμα της ρύθμισης επίσης των κρατικών επιδοτήσεων, των κρατικών ενισχύσεων. Δεύτερο σημείο, συμπίπτω απόλυτα με εκείνους που ανέφεραν πιο πριν <clears throat> ότι είναι τεράστια η σημασία αν θέλουμε να εμβαθύνουμε στην ενιαία εσωτερική αγορά και τη δημιουργία της, να προχωρήσουμε, αν θέλουμε να προχωρήσουμε προς μια ενεργειακή πολιτική μιας κοινή αγοράς ενέργειας και ενεργειακών πόρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε στις διασυνδέσεις. Και αυτό είναι ένα σημείο το οποίο δεν έχουμε επιλύσει μέχρι σήμερα. Σημειώνονται πρόοδοι, σημειώνονται δηλώσεις που έχουμε, διακηρύξεις προθέσεων που λένε ότι θα πρέπει να υπάρξουν περαιτέρω πρόδια, αλλά δεν έχουμε επιλύσει τη διασύνδεση. Και δεν την έχουμε επιλύσει επειδή είναι πολύ δύσκολο θέμα. Ακαθόδες από ένα ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο να ρυθμιστεί και να αντιμετωπιστεί εδώ στις Βρυξέλλες. Να ξεπεράσουμε όλα τα προσκόμματα και τα εμπόδια τα οποία δημιουργούνται λόγω των αντιφατικών συγκρουόμενων συμφερόντων κάποιων κρατών μελών έναντι των συμφερόντων άλλων κρατών μελών. Όταν έρχεται η ώρα να θέσουμε την εκμετάλλευση των πόρων με τη βούλησή μας από κοινού και να οικοδομήσουμε και να γίνει λειτουργική μια τέτοια διασύνδεση. Έχουμε βελτιώσει με την μορφή και τον τύπο των συντονιστών σχεδίων διευρωπαϊκών προγραμμάτων και δικτύων, αλλά δεν έχουμε επιλύσει όλα τα προβλήματα. Σίγουρα υπάρχουν περισσότερα προβλήματα και πρέπει να συνεχίσουμε να τα εξετάζουμε. Ένα από αυτά και δεν είναι το μικρότερο και δεν είναι το μόνο, <clears throat> είναι η χρηματοδότηση σίγουρα. Οι χώρες, τα κράτη-μέλη λένε όταν και αν πρόκειται να γίνει μια επένδυση για να διασυνδεθούν τα δίκτυά μας με τα δίκτυα άλλων χωρών, να το πληρώσει λέει η Ευρώπη αυτό ως χρηματοδότηση. Όχι εμείς λένε αυτοί, η Ευρώπη να τα χρηματοδοτήσει. Και αν πάτε εσείς να αναλύσετε τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και δείτε που αποφασίζετε εδώ σε αυτό το Ευρωκοινοβούλιο σε διάλογο με τις κυβερνήσεις, τις εθνικές κυβερνήσεις προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. όμω η Δημοσιονομική Αρχή που είναι αυτή εδώ η Εθνική Βουλή, το, με συγχωρείτε το, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη-μέλη που ενώνονται στο Συμβούλιο, θα δείτε δεν υπάρχουν επαρκή κονδύλια. Βρισκόμαστε πολύ μακριά. Πόρο απέχουμε από το να μπορέσουμε να εντάξουμε στον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό τα κονδύλια που θα ήταν αναγκαία να ενταχθούν σε αυτόν και να εγγραφούν σε αυτόν για να χρηματοδοτήσουμε από τον κοινοτικό προπολογισμό αυτά τα εγχειρήματα και τα σχέδια κοινοτικού Έχουμε άλλο μέσο χρηματοδοτικό που συνεργάζεται για τη συγχρηματοδότηση. Ένα καθαρά ευρωπαϊκό μέσο που είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η ΕΤΕ. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων κάνει μεγάλη προσπάθεια για να χρηματοδοτήσει και να χρηματοδοτηθούν με, τους, με τα κονδύλια, με τους πόρους που αντλεί από τις αγορές αυτά τα εγχειρήματα. Αλλά έχει όρια, έχει περιορισμούς και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Έχει περιορισμένη ικανότητα χρηματοδότησης, γιατί. Λόγω των μετόχων, όπως κάθε τράπεζα έχει τους μετόχους. Ποιοι είναι οι μέτοχοι <laughs> της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, τα κράτη-μέλη είναι οι μέτοχοι. Εκείνοι αποφασίζουν τι είναι εκείνο το οποίο μπορεί ή δεν μπορεί να χρηματοδοτήσει η ΕΤΕ, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Λοιπόν, για αυτούς τους λόγους υπάρχουν χρηματοδοτικά προβλήματα πάρα πολύ σημαντικά, τα οποία ποτέ δεν θα μπορέσει να επιλύσει μόνο και αποκλειστικά ο δημόσιος τομέας των κρατών μελών ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να πετύχουμε να αντλήσουμε κονδύλια κονδύλια, κεφάλαια από τον ιδιωτικό τομέα. Και δεν είναι αυτή ακριβώς η καλύτερη και πιο εύκολη χρονική στιγμή, η πιο κατάλληλη και ευνοϊκή χρονική στιγμή για να αντλήσουμε κονδύλια από τον ιδιωτικό τομέα. Αλλά με μια προοπτική στο μέλλον, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, από εκεί πρέπει να δοθεί η λύση. Μεγαλύτερη ικανότητα πολιτική να ξεπεράσουμε τα προβλήματα και τα προσκόμματα. Μεγαλύτερη χρηματοδοτική ικανότητα. Μοχλεύοντας και αυξάνοντας πολλαπλασιαστικά την ικανότητα των κονδυλίων του ευρωπαϊκού προπολογισμού με τα κονδύλια τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, συν επιπλέον τα κονδύλια του ιδιωτικού τομέα που θα συνεισφέρουν. Και όπω πάντα, μεγαλύτερη πολιτική υποστήριξη ώστε όλα αυτά να είναι εφικτό να ενταχθούν σε μια συνεκτική ενιαία πολιτική. Τώρα, για το θέμα των τεχνολογιών. Αναφέρθηκαν λογικά πράγματα με τα οποία συμφωνώ ο Πέντρο Μαρίν. Ένα μόνο σχόλιο έχω να κάνω. Επειδή υπήρξαν κάποιες παρεμβάσεις σε σχέση με τον τομέα των αυτοκινητοβιομηχανιών ή γενικότερα των πολιτικών της μείωσης και της, ε, των εκπομπών ρήπων. Προσπαθώντας να εντάξουμε και να το ε, ε, εντοπίσουμε σε αυτές τις πρωτοβουλίες μια ευρύτερη πρωτοβουλία. Δεν είναι μόνο αυτά τα οποία πρέπει να γίνουν. Είναι σαφές ότι δεν είναι, είναι προφανές ότι αυτές δεν είναι οι μόνες προσπάθειες που πρέπει να γίνουν. Αλλά είναι οι προσπάθειες που είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε. Υπάρχουν περισσότερα πράγματα να κάνουμε. Αλλά αν δεν κάνουμε μία φιλόδοξη πολιτική και αποτελεσματική ταυτόχρονα ελέγχου εκπομπών ρήπων διοξιδίου του άνθρακα, εντάσσοντας και χρησιμοποιώντας όλα τα αναγκαία μέσα και μέτρα στην εξυπηρέτηση των στόχων που θέσαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και που έχουμε ενώπιόν μας ως διεθνής κοινότητα, τότε θα κάνουμε ένα τεράστιο σφάλμα. Όχι μόνο τεράστιο σφάλμα <clears throat> μη έκφρασης αλληλεγγύης για τις επόμενες γενναίες και τον πλανήτη μας, την οικουμένη μας, αλλά τεράστιο σφάλμα υπό το πρίσμα και οικονομικής δράσης η καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών, οι νέε πιο αποτελεσματικέ τεχνολογίε για τον ενεργειακό τομέα κτλ. κτλ Αυτοκινητοβιομηχανίε κτλ. Όλα αυτά είναι ένα από του κύριου μοχλού για να διαφύγουμε από τη σημερινή κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε και να αντιμετωπίσουμε την μικρή παραγωγικότητα και μικρή ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να αντέξουμε και να αυξήσουμε τους ρυθμούς στην οικονομική ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα. Και να μην υποβάλουμε, να μην ε, υπάρξει σε σχέση με τους ανταγωνιστές μας άλλες χώρες και άλλους, ε, είπα για παράδειγμα, <clears throat> η υποχρεωτική αυτή ε, πτυχή της απεμπόλησης ε, της ε, κλιματικής συνιστώσας ε, και της καταπολέμησης των κλιματικών αλλαγών και για τις κυριότερες αναδυόμενες τεχνολογίες, ε, οικονομίες. Είναι ένα καθαρά και καθαρά οικονομικό συμφέρον που πρέπει να μας κάνει να δούμε ότι οι κλιματικές αλλαγές και η καταπολέμησή τους πρέπει να είναι μία από τις μεγαλύτερες προτεραιότητες μας. Όχι μόνο υπό τον ενεργειακό τομέα και πρίσμα, αλλά και υπό την σφαιρικότερη δράση και πολιτική μας. Και δύο σύντομα σχόλια για τις εθνικές ιδιομορφίες και τη σημερινή συνθήκη και κατάσταση των πραγμάτων. Είναι σαφές ότι υπάρχουν πολλές εθνικές ιδιομορφίες και είναι σεβαστές αυτές. Για παράδειγμα, η συζήτηση που ξεκίνησε και άνοιξε με διάφορες, διαφορετικές παρεμβάσεις που απέρευσαν από το ημικύκλιο εδώ, την Ολομέλεια, για την πυρηνική ενέργεια, ανανεώσιμες ε, πηγές ενέργειας, μίξ ενεργειακό, ενεργειακό μείγμα. Θα συνεχιστεί αυτή η συζήτηση, διότι δεν υπάρχει μία και μόνο ε, αναδυόμενη ευρωπαϊκή πολιτική στον άμεσο χρονορίζοντα. Είναι θέμα της κάθε χώρας μέλος. Και βάση αυτή τη αρμοδιότητα κάθε κράτο μέλο να αποφασίζει το κάθε κράτο μέλο για αυτό το μείγμα το ενεργειακό το οποίο χρειάζεται, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δημιουργήσει μια ενιαία ενεργειακή αγορά στην Ευρώπη και μια στρατηγική που θα υιοθετήσει για την καταπολέμηση των ε, ε, κλιματικών αλλαγών που θα είναι κοινή. Είναι αυτό δύσκολο να γίνει σε σχέση με την επιλογή ενός ενεργειακού μίξ, αλλά αυτό είναι το στίχημα, το διακύβευμα το οποίο έχουμε ενώπιόν μας. Μια άλλη πτυχή των εθνικών ιδιομορφιών στις οποίες αναφέρθηκαν κάποιοι από εσά είναι τα θέματα φορολογίας. <clears throat> Στα ενεργειακά θέματα υπάρχουν ειδικοί ε, δασμοί και τέλη. Υπάρχουν οδηγίες που θέτουν σε ευρωπαϊκή είναι επίπεδο ένα ελάχιστο επίπεδο εσόδων ή τελών για, τα, για τους υδρογονάνθρακες. Δεν υπάρχει όμως ένα εναρμονισμένο σύστημα. Συζητάμε μια νέα οδηγία τώρα για το ενεργειακό κόστος που θα πρέπει να μπορεί να καλύπτεται. Ακόμα δεν έχει υποβάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια τέτοια πρωτοβουλία ως πρόταση, αλλά θα το κάνει σύντομα. Προσπαθούμε μέσα από αυτά τα τέλη να διαφοροποιήσουμε για ποια ενέργεια κάνουμε λόγο για τη συνιστόσα την ενεργειακή και την περιβαλλοντική συνιστόσα. Ε, εργαζόμαστε προς αυτή την κατεύθυνση και γίνονται συζητήσεις σε κάποια κράτη-μέλη αλλά επίσης και σε κλίμακα Ευρωπαϊκής Ένωσης γίνονται συζητήσεις για τη δυνατότητα εισαγωγής ενός τέλους ε, για τον άνθρακα. τέλο που θα επιβαρύνει τον άνθρακα. Που προσωπικά εγώ ίδιο πιστεύω ότι είναι μια καλή κατεύθυνση που μπορούμε να ακολουθήσουμε. Αλλά ακόμα δεν είναι μια πορεία που να βασίζεται στην υποστήριξη όλων των κρατών μελών. <clears throat> εδώ εξαιρείται η Σουηδία η οποία έχει εδώ και χρόνια ένα τέτοιο τέλος επί του άνθρακα αλλά το συζητάμε τώρα ως προοπτική σε ευρωπαϊκή κλίμακα. Η Ευρατόμ θέτει και την κλίμακα για τα ότι σε σχέση με τα κονδύλια τα οποία διατίθενται είναι ε, θέματα ασφάλειας μόνο. Δεν είναι η ανάπτυξη της πυρηνικής ενέργειας, είναι η κάλυψη της συνιστώσας μόνο της ασφάλειας των ε, πυρηνικών αυτών συνιστώσεων. Και τέλος η συνθήκη τη Λισαβόνα. Συζητώντα αν επαρκεί η συνθήκη τη Λισαβόνα ή όχι, είναι ένα σκόπιμο ερώτημα, αλλά που τίθεται υπερβολικά νωρί. Είναι πολύ πρόημο. Ακόμα τώρα, καλύτερο είναι να απαντήσουμε ερωτήματα γιατί δεν κάναμε όλα όσα μπορούσαμε να κάνουμε πριν από τη συνθήκη τη Λισαβόνα. Και ιδιαίτερα όπως είπα στην αρχή κιόλας και είπαν και κάποιοι από εσά ε, στις παρεμβάσεις σας, να μεταφέρουμε σε κάθε μία από τις νομοθετικές τάξεις των κρατών μελών μέχρι το Μάρτιο του 2011 το τρίτο πακέτο όσον αφορά τα νομοθετικά μέτρα που λάβαμε. Να μεταφερθούν και να υλοποιηθούν αυτά στα κράτη-μέλη. Πολύ σημαντικό αυτό. Μετά πρέπει αυτά παράλληλα να αναπτύξουν, να αναπτύξουν αυτά τα οποία προβλέπονται στην στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα μέτρα για το 2020. Αντιμετώπιση κλιματικών αλλαγών να αναπτυχθεί μια νέα νομική βάση από τη συνθήκη τη Λισαβόνα που μόλι άρχισε να ισχύει. Πράγμα που δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να συζητήσουμε με μια προοπτική προ το μέλλον, με ένα ε, όραμα πιο μακροπρόθεσμο για το τι πρέπει να κάνουμε επιπλέον. Πέρα από εκείνα τα οποία υποχρεωτικά πρέπει να κάνουμε αυτού του μήνε ή στα επόμενα δύο χρόνια υποχρεωτικά. Είναι αυτονόητο ότι πρέπει να μπορέσουμε να συζητήσουμε με ένα όραμα και προσέγγιση μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο. Αλλά η προσωπική μου σύσταση είναι να συζητήσουμε πρώτα επί της ουσίας, επί των θεμάτων ουσίας και μετά να καλέσουμε ε, καθηγητές συνταγματικού δικαίου να μας πούν πώς μπορούμε να πετύχουμε αυτά τα οποία επιθυμούμε να πράξουμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επί πολλά χρόνια δυστυχώς <clears throat> αφαιρούσε, αν μου επιτρέπετε, συγγνώμη για όσους βρίσκονται εδώ, έδινε υπερβολική προσοχή στα συνταγματικά θέματα και υπερβολικά λίγη προσοχή στις Φιλοδοξίε τις πολιτικέ ε, για να συνεχίσουμε την οικοδόμηση τη Ευρώπη. Αυτή είναι η προσωπική μου εντύπωση. Και εγώ πιστεύω ότι τώρα πρέπει να τεθούν τα πράγματα στη σωστή σειρά και αλληλουχία. Πρώτον, τι θέλουμε να κάνουμε, γιατί και πώ και ποιο κατεπήγον χαρακτήρα υπάρχει στην υλοποίησή του και μετά να διαρωτηθούμε ποιε είναι οι νομικέ εκείνε μεταβολέ και τροποποιήσει που χρειάζονται ε, και που, για να πετύχουμε αυτά που θέλουμε. Μεταξύ άλλων ε, θεμάτων, πριν καλέσουμε έναν καθηγητή συνταγματικού δικαίου θα πρέπει να δούμε τι πρέπει να ρυθμίζονται από τα δημοσιονομικά στο ευρωπαϊκό επίπεδο για τις, προοπτικές, τις μελλοντικές προοπτικές 2014-2020 και να δούμε τι πρέπει να γίνει και γιατί δεν μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε λόγω έλλειψης κονδυλίων ε, ε τις αναγκαίε ευρωπαϊκές Είναι μια συνέχεια της συζήτηση που πρέπει να γίνει και τι ανάγκε να δούμε μετά για την αλλαγή νομικών βάσεων. Ευχαριστώ. Κύριε Αντιπρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, βέβαια συνεχίζουμε αυτό ήταν ε, μία περίληψη της συζητήσεως. Η συζήτηση αυτή ε, ξεκίνησε πριν από λίγες εβδομάδες και αυτός ήταν μόνο ένα σταθμό στη συζήτηση. Ίσως ε, αυτές οι ενέργειες είναι πιο εύκολο να εφαρμοστούν σε περίοδο κρίσεως γιατί ξέρουμε αυτή τη στιγμή και είναι προφανές για όλους μας πόσο σημαντικό είναι να ολοκληρώσουμε την εσωτερική αγορά που αποτελεί ένα από τα βασικά θέματα. Και ένα από τα βασικά αυτά θέματα είναι η ενεργειακή αγορά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και την ε, Ισπανική Προεδρία για μια τόσο σημαντική προτεραιότητα. Την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία προτείνει μια, ε, ένα πρόγραμμα δράσεως ε, για το 2020. Ευχαριστώ κύριε Αντιπρόεδρε επίσης διότι αναφέρεστε σε πολλά θέματα. Βεβαίως θα, θα έρθω σε επαφή με τον κύριο Ζακ Ντελόρ, πρώην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μόνο την Επιτροπή για να ετοιμάσουμε τις πρώτες απαντήσεις μας. Τι είναι βασικό. Ορισμένα θέματα νομίζω ότι την χάνουν γενική συνένεση μεταξύ μας. Εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα πρώτο βασικό σημείο. Δίκτυα για την ενέργεια ε, αντίδραση στις κρίσεις, ε, θέμα έρευνας. Ε, έχουμε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα ε, για την ενέργεια, στρατηγική του 2020. Πώς θα μπορέσουμε να εφαρμόσουμε τα προγράμματά μας στη στρατηγική και από πλευράς προϋπολογισμού. Επίσης η χρήση της, της ενέργειας είναι ένα θέμα αλλά οι ανανεώσιμες ενέργειες είναι ένα άλλο και πόσο θα μπορέσουμε να μειώσουμε τις εκπομπές της ενέργειας είναι ένα άλλο διότι στην Κίνα παραδείγματο χάρη δεν θέλουν ε, να αλλάξουν και να εγκαταλείψουν ε, τους ενεργειακούς ε, σταθμούς που χρησιμοποιούν άνθρακα κατά 40% ενώ εμείς έχουμε 14% μόνο. Επίσης το θέμα CCS, Carbon Capture and Storage, είναι πολύ σημαντική τεχνολογία. Πρόκειται για τη δέσμευση και την αποθήκευση του διοξιδίου του άνθρακος. Ε, βεβαίως χρειάζονται κίνητρα για τις εταιρείε μας. Πρέπει να είναι ανταγωνιστικές θα θέλανε να αρθούν τα εμπόδια, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και επίσης το θέμα του κόστους της ενέργειας, της τιμής της ενέργειας, πολύ βασικό για τους πολίτες και για την ανταγωνιστικότητα όλης της οικονομίας. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να σας πω και να δούμε πώς μπορούμε να επιλύσουμε νομικά το θέμα αυτό ε, αυτό θα είναι το θέμα της επόμενης συζήτησής μας, δηλαδή τα κράτη-μέλη θα πρέπει να αποφασίσουν τελικά εάν θέλουν ή όχι να συμμετάσχουν σε αυτήν την κοινή πολιτική ή στην ε, ε, κοινοτική πολιτική ενεργείας. Ε, πολιτική ορμή. Νομίζω ότι όλοι αναφερθήκατε σε αυτό και νομίζω ότι η πολιτική βούληση είναι και εδώ σήμερα. Τα εθνικά κοινοβούλια είναι πολύ σημαντικά. Μπορούμε να ξεκινήσουμε μια τέτοια συζήτηση στα εθνικά κοινοβούλια μας εάν εσείς το αποφασίσετε και επιλέξετε να το πράξετε, ε, όπως γίνεται και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εμείς από τις αρχές Μαΐου έχουμε ξεκινήσει αυτή τη συζήτηση, οπότε δεν, ε, δεν προπορευόμαστε πάρα πολύ ε, χρονικά από σας. Σας ευχαριστώ όλους για την παρουσία σας εδώ. Ευχαριστώ όλους όσους συμμετείχαν εις ε, την οργάνωση και θα ήθελα να προσθέσω ότι όλα τα στοιχεία της ε, κοινής συνεδριάσεώς μας όσον αφορά την ενέργεια βρίσκονται στο διαδίκτυο ή στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου europarl.europa.eu ε, Έχετε ε, έγγραφα και έξω από την αίθουσα τα οποία μπορείτε να πάρετε. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ για την εξαιρετική συζήτηση και η επόμενη συζήτηση θα οργανωθεί ίσως ή στα εθνικά σας κοινοβούλια ή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι κάτι το οποίο θα σκεφτούμε. Σας ευχαριστώ όλους.